για την γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος για πρότυπα για τις επιδόσεις καινούριων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων όσον αφορά τις εκπομπές. Η πρώτη ψηφοφορία είναι η συμβαστική τροπολογία Α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Μετά έχουμε την Β. Δεν ξέρω, τρία αναφέρεται στο δικό μου κατάλογο. Β, υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 43 κύριε Στέρξ υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική γάμα υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσουμε την γάμα αρχιτή ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. 17 υπέρ 16 κατά δύο αποχές. Γίνεται λοιπόν δεκτή η συμβαστική γάμα. Μετά έχουμε τις τροπολογίες επί των ημερομηνιών που ξεκινάνε στο άρθρο 7 παράγραφος 1. Οπότε θα ψηφίσουμε unblock 16 νομίζω τροπολογίες. Α, όχι, ψηφίσουμε το block 16, συγγνώμη. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. μεταψίζουμε το μπλοκ 17 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ να ελέγχουμε το μπλοκ 17 έρχεται ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας 17 υπέρ 18 κατά απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία δέλτα υπέρ κατά αποχές δεκτή ε υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσουμε την ε και αρχιτεί ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας 17 υπέρ 18 κατά απορρίπτεται 95 της κυρίας Βουίλς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 94 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε την 94 αρχιτεί ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρασε 17 υπέρ 17 κατά μία αποχή απορρίπτεται μετά έχουμε την 101 Ναι, 101 καλύπτεται από το 95, οπότε περνάμε στην 100 του κυρίου Ελχαντραγουή υπέρ. Κατά αποχές θα επαληθεύσουμε την 100 του κυρίου Ελχαντραγουή. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρασε. 19 υπέρ, 16 κατά, γίνεται δεκτή. Παίρναμε λοιπόν στην 126 υπέρ, κατά αποχές. Να επαληθεύσουμε την 126 παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρας 18 υπέρ 17 κατά δεκτή 50 ελ χαντραουί υπέρ κατά επαληθεύσουμε την 50 του κυρίου Ελχαντραουή άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 18 υπέρ, 17 κατά καμία εποχή. Ο κύριος Τέιλορ θα σκέφτεται πω, πω, πω όλα τσιμα τσιμα είναι. Τόσο δεν είναι πάντα όλες έτσι ε, οι ψηφοφορίες. Περνάμε στην επόμενη, την 52 υπέρ. Νομίζω το έλκει είναι κατά. Κατά. Αποχές θα επαληθεύσουμε την 52 αρχιτή ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 18 υπέρ 17 κατά γίνεται δεκτή. 51 καταπίπτει. Οπότε ψηφίζουμε το μπλοκ 18. Κοιτάξτε, κάποιοι λένε ότι όταν ξεκινήσει η ψηφοφορία δεν κάνει να μπαίνει κανεί μετά, αλλά δεν θα το τραβήξω τόσο. Λοιπόν, ψηφίζουμε το μπλοκ 18 υπέρ κατά αποχές θα το επαληθεύσουμε ψηφίζουμε λοιπόν το μπλοκ 18 να δούμε τι θα αλλάξει με τον κύριο Φιντέντσα. Άρχεται η ψηφοφορία. As everybody voted. Ψήφισαν όλοι. All abuse of the chair. The vote is closed πέρας της ψηφοφορίας βλέπετε κάνω κατάχρηση της θέσης μου. Αλλά δεν είχε καμία σημασία, 24 υπέρ 13 κατά. Περνάμε στην 68. Ο κύριος Φιντάντσα ήρθε βεβαίως στην ώρα για να ψηφίσει τη δική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 70 Οπότε ψηφίζουμε την 87 μου λένε εδώ πέρα η υποβολής του κυρίου Λιμπεράτσκι λοιπόν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 109 της κυρίας τικα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. καταπίπτουν. Περνάμε λοιπόν στροπολογίες του pooling για τους κατασκευαστές. Unblock από την 88 μέχρι την 104 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στις υπόλοιπες τροπολογίες. 55 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση της 55 άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. 18 υπέρ 18 κατά απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές δεκτή 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καταπίπτει 89 Τις επόμενες τις ψηφίζουμε αν μπλόκα 90 με 99. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 90 με 99. 90, 96, 97, 98, 99. Ψήφισαν όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. 18 υπέρ, εγκρίνεται. 35 υπέρ, συγγνώμη, εγκρίνεται. Η 110 καταπίπτει, 111 της κυρίας Φαγιών, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 127, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 17 του εισηγητού. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 132 της κυρίας Τικάου. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 18 του εισηγητού. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 134 υπέρ, κατά, αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε για την 134. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Ναι. Πέρα στις ψηφοφορίες. 19 υπέρ, 19 κατά, απορρίπτεται. 136 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 138 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 140 υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω ότι απορρίφθηκε, αλλά θα το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 140. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 18 υπέρ, 20 κατά, απορρίπτεται. 150. Ποιοι είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω ότι απορρίφθηκε, αλλά θα το ελέγξουμε. Έλεγχος για την 151 αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας, 15 υπέρ, 23 κατά, απορρίπτεται. 24 χωριστή ψηφοφορία εδώ. Πρώτη παράγραφος, ποιοι είναι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερη παράγραφος, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε και αυτή. 152 του κύριου Ταταρέλα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε την 152 και την 153. Είναι ταυτόσιμες. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 18 υπέρ, 20 κατά. Απορρίπτεται. 154 και 155. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται. 162. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 166. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 32 η επόμενη. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 41 καταπίπτει λόγω της συμβιβασμού Β. 44. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49. Καταπίπτει. Και έτσι περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. 32 υπέρ, 40 κατά, 2 αποχές. Επομένως εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Βλάσακ. Συνάδελφοι, επειδή είστε τόσο αποτελεσματικοί και επιθαρχημένοι, έχουμε την Επίτροπο Δαμανάκη, η οποία θα έρθει στις 10 παρατέταρτο και γι' αυτό πρέπει να αναστείλουμε τις εργασίες μας μέχρι την άφηξη της Επιτρόπου. Σας παρακαλώ λοιπόν μην απομακρυνθείτε πολύ για να ακούσουμε την Επίτροπο και φυσικά και η κυρία Μάισνερ μπορεί να την ε, σταυρώσει με μεγάλη ζέση. Λοιπόν, στις 9 παρατέταρτο. Στις 10 παρατέταρτο. Okay, colleagues. I don't know whether... Εντάξει, συνάδελφοι, δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια μέλη της Επιτροπής μας έξω. Παρακαλώ, αν υπάρχουν κάποια έξω, φωνάξτε τους μέσα. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, λοιπόν, είναι η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Η συγγήτρια είναι η κυρία Μάισνερ. αλλά με μεγάλη μου χαρά καλωσορίζω την Επίτροπο, την κυρία Δαμανάκη, στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού σήμερα το πρωί. Έχουμε ένα είδος διαρκούς συνεννόησης με την, Ευρωπα... με την Επίτροπο, Αντιπρόεδρος Κάλλας, έχουμε τον κύριο Ταγιάννη στον τουρισμό στο, εν τέλει γνωρίζουμε πολύ καλά τους επιτρόπους μας στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Σας καλωσορίζουμε σήμερα εδώ και σας εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας που ήρθατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση. Αν θέλετε να λάβετε το λόγο, είμαι βέβαιος ότι τα μέλη και η κυρία Μάισνερ θα έχουν πολλά πράγματα να πούν μετά από την παρέμβασή σας. Έχετε το λόγο, κυρία Επίτροπε. Very much, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ. Υπόσχομαι να μην πω στα χωράφια του κύριου Ταγιάννη και Κάλλας. Ε, κύριε Πρόεδρε, κυρία Μάισνερ, ε, αγαπητά μέλη, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχήν για την ευγενική σας πρόσκληση πάνω στο σχέδιο έκθεσης ε, για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της κυρίας Μάισνερ. Αυτή η έκθεση δεν είναι μια απλή έκθεση καταγραφής. Ανα... Αναθεωρεί την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμετοχή σας επιβεβαιώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση του Κοινοβουλίου μας. Είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Σήμερα περισσότερο από ποτέ τα συγκεκριμένα ωφέλη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στα θαλάσσια πράγματα είναι επίκαιρη όσο ποτέ. Η πετρελαιοκυλίδα στο Μεξικό, η ταχύτατη εξάπλωση της πειρατείας είναι μόνο δύο παραδείγματα που έφτασαν στις εφημερίδες. Υπάρχουν παραδείγματα πολύ μεγαλύτερων δικτύων προκλήσεων. Οι πιέσεις που δέχεται το θαλάσσιο περιβάλλον, η απώλεια βιοπικιλότητας, η αλλαγή του κλίματος, η αυξημένη εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων, συμπεριλαμβάνει της υπεραλίευσης φυσικά, ε, τρέχουν παράλληλα και δημιουργούν μια πρόκληση που είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των μερών της. Επίτσι, η προσέγγιση μας πρέπει να βασίζεται σε μια συνεκτική θεώρηση η οποία διατρέχει όλες τις πολιτικές. Αυτή είναι η ουσία μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής στο κάτω-κάτω. Να υπάρχουν θετικές δράσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ όλων των πολιτικών και των κοινωνικών συμφερόντων, προσπαθώντας να συνδυάσει τις προσπάθειες από όλους τους τομείς για την αύξηση της αποτελεσματικότητας. Αλλά εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, Επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια για τις διαφορετικές προτεραιότητες τις οποίες υπηρετώ από τότε που ανέλαβα τα αξιώμα μου το περασμένο Φεβρουάριο. Ας ξεκινήσω με, το, με την Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 για τον βιώσιμη ανάπτυξη, την οικονομική μεγέθυνση και την ανάπτυξη της απασχόλησης. Πιστεύω σταθερά ότι οι διάφοροι θαλάσσιοι τομείς μπορούν να προσφέρουν και να συμβάλλουν πολλά, ιδίως αυτούς τους δύσκολους οικονομικούς καιρούς. Τον περασμένο μήνα απευθύναμε μια έκκληση για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη, μια μελέτη. Η μελέτη αυτή θα μας φέρει πιο κοντά στον στόχο μας μιας διατομεακής προσέγγισης για τη βιώσιμη πολιτική στις παράκτιες ζώνες και στις θαλάσσιες περιοχές για την, τα παραδοσιακά θαλάσσια επαγγέλματα όπως η αλληλείς και η ναυτική για τους, οποίους, για τους οποίους θα ήθελα να εξασφαλίσω στα διαδρομίες αλλά και για τα νέα επαγγέλματα τα οποία θα αναδυθούν από τους νέους θαλάσσιους τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές και οι γαλάζιες βιοτεχνολογίες. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης θα τα έχουμε το 2012. Μια άλλη προτεραιότητα είναι να συνδυάσουμε την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος με την ανάπτυξη των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό εξερευνώντας τα όρια της, της βιωσιμότητας όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που έχουν επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτό έχει πολλές πρακτικές επιπτώσεις για την οδηγία για τη σχετική οδηγία και για το πακέτο για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια. Η τρίτη προτεραιότητα έχει να κάνει με τις στρατηγικές του θαλάσσιου πυθμένα. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες προτεραιότητες οι οποίες προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες. Ανάλογα με τις πολιτικές, πολιτικοκοινωνικές και φυσικές παραμέτρους. Πρέπει επίσης να δούμε τις ιδιομορφίες των διαφόρων περιοχών από την Αρκτική, τη Βαλτική μέχρι τη Μεσόγειο. Με βάση τα συμπεράσματα του τελευταίου Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής θα παρουσιάσουμε μια νέα στρατηγική για τον Ατλαντικό μέχρι τον Ιούνιο του 2011. Μια τέταρτη προτεραιότητα έχει να κάνει με τα διάφορα εργαλεία τα συστήματα επιτήρησης, τη δικτύωση των θαλάσσιων δεδομένων. Η εργασία πάνω στα εργαλεία αυτά έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Σκοπεύουμε να εκδώσουμε μια ανακοίνωση για την θαλάσσια χωροταξική πολιτική πριν από το τέλος αυτού του έτους και θα παρουσιάσουμε νομοθετικές επιλογές για τη διαμόρφωση μιας κοινή προσέγγισης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο για την ολοκλήρωση της θαλάσσιας επιτήρησης, συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για να προτείνουμε μέχρι τον επόμενο Οκτώβριο, δηλαδή το 2010, έναν οδικό χάρτη προς την εγκαθίδρυση ενός κοινού περιβάλλοντος ε, διαμήρασης πληροφοριών και δεδομένων. Αυτό θα επιτρέψει τις εθνικές αρχές ε, σε όλες τις θαλάσσιες δραστηριότητές τους, είτε αυτή είναι η καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης, η καταπολέμηση άλλων παράνομων δραστηριοτήτων ή και η διεξαγωγή νόμιμων δραστηριοτήτων. Το τέταρτο γεύμα, ε, η, συγγνώμη, ο θαλάσσιος Άτλαντας που θα δημοσιευθεί, θα διευκολύνει τη ζωή όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Θα είναι μια ανακοίνωση που θα εμβαθύνει τις γνώσεις όλων των πολιτών της Ευρώπης. Πέμπτον, το να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια διεθνή διάσταση στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Θα πρέπει εδώ πέρα να επιμείνουμε στον ηγετικό ρόλο που μπορεί να δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την θαλάσσια διακυβέρνηση. Θέλουμε να κυρωθεί η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Επίσης πρέπει να συνεχίσουμε την εργασία μας προκειμένου να πετύχουμε έναν καλύτερο ρόλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε διεθνή φόρα όπως ο Διεθνής Οργανισμός για την Θάλασσα. Θέλουμε βέβαια επίσης να έχουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση και τα απαραίτητα σχετικά μέσα για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Μετά το καλοκαίρι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει ένα σχέδιο κανονισμού για τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένη θαλάσσης πολιτικής για τα επόμενα δύο χρόνια προτείνουμε 50 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2011 και 2012 βάσει των ποσών που έχετε ήδη εσείς δώσει στην προπαρασκευαστική φάση. Ε, παθιόμαστε λοιπόν στη δική σας υποστήριξη προκειμένου να αρχίσει να ισχύει ο κανονισμός αυτός το 2011 και προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι η νέα ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική θα έχει τον κατάλληλο ρόλο που πρέπει να κατέχει στα πλαίσια των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω ότι η εργασία της Επιτροπής σας εμπνέεται από ένα γενικότερο πνεύμα συνεργασίας. Το να συνεργαστούμε λοιπόν μαζί για διάφορες πολιτικές θα μας επιτρέψει να εντοπίσουμε τις συνέργειες που μπορούμε να έχουμε και θα καταφέρουμε να πετύχουμε την απαραίτητη συνεργασία που απαιτεί ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Ξέρετε ότι ε, η θάλασσα είναι ένας παράγοντας που μας συνώνει όλους και μας γεμίζει με ελπίδα. Και η φράση αυτή παίρνει μια, ένα άλλο νόημα αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο πλοίο, στο ίδιο σκάφος και ξέρω ότι στα πλαίσια της Επιτροπής αυτής θα έχω ένα πραγματικό συνεργάτη, ένα πραγματικό εταίρο και συνομιλητή προκειμένου να κινηθεί το πλοίο αυτό σωστή κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Όπως περιμένετε υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κατάλογος ομιλητών. Θα ξεκινήσουμε με την εισηγήτριά μας, την κυρία Μάισνερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε για τα λόγια τα οποία είπατε. Όντως, έγινε μια συζήτηση για το ζήτημα αυτό της ολοκληρωμένης θαλάσσης πολιτικής και με έχει απασχολήσει πάρα πολύ ακόμα και προσωπικά. 320.000 χιλιόμετρα ακτές έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα πολύ μεγάλο τμήμα του ευρωπαϊκού πληθυσμού εξαρτάται από το θαλάσσιο περιβάλλον. Ακόμα και άνθρωποι που ζουν στην ενδοχώρα επηρεάζονται από την ε, οικονομική ανάπτυξη των ε, παράκτων περιοχών και ένα 40% του ε, ευρωπαϊκού ΑΕΠ προέρχεται από τις περιοχές αυτές. Είναι λοιπόν προφανές ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στις απαραίτητες προτάσεις που θα έχουν κυρίως να κάνουν με τις ε, μεταφορές και με την καλύτερη διασύνδεση της ενδοχώρας με τις παράκτιες περιοχές. Επομένως... Κοιτάξτε, δεν ε, προσφέρει τίποτα να αναπτύσσεται ο ένας τομένας ε, χωριστά από τον άλλο στο μέλλον. Θα πρέπει όλοι αυτοί να πάνε μαζί και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συμβάσουμε αυτούς τους τομείς στη μελλοντική μας ε, εργασία και την αυτιλία και τον τουρισμό και την υπεράκτια ενέργεια και την αλληλεία και την προστασία των ακτών και τη θαλάσσια οικολογία και την επιτήρηση των ακτών, τη θαλάσσια έρευνα με την ε, γαλάζια τη λεγόμενη βιοτεχνολογία και όλα αυτά βέβαια υπό την επίδραση της προστασίας του κλίματος. Και βεβαίως ε, βλέπουμε πως ε, δεν ξέρω ε, εκεί που προγραμματίζονται ταυτόχρονα νέα αυτοκινητόδρομοι θα ε, βλέπουμε πως θα μπορούσαν να αναπτυχθούν νέες υπεράκτιες τοποθετήσεις ΑΠΕ και ταυτόχρονα να υπάρχει και τα δραστηριότητα αλίας και όλα αυτά να συμβάζονται και ίσως να δούμε πώς έτσι θα αναπτυχθούν και περισσότερες θέσεις εργασίας. Νομίζω και ο στόχος για την Ευρώπη 2020 θα υποφεληθεί από αυτή την προσέγγιση. Αν προσπαθήσουμε λοιπόν να αποφύγουμε την αλληλεπικάλυψη, τους διαφορούς καυγάδες και να υπάρχει ένας κοινός προγραμματισμός. Αυτό γίνεται στην κοινή θαλάσσια πολιτική και βλέπω πως ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να απασχολούνται από αυτά τα πράγματα γιατί απασχολούνται σε τομεί που σχετίζονται με την θάλασσα, δεν τα γνωρίζουν πλήρω αυτά τα πράγματα. Ένα στόχο που έχω είναι αυτό, να γίνει γνωστό αυτό το πράγμα και με καθοδήγησε αυτό η σύνταξη τη έκθεσή μου. Γνωρίζετε πω ε, έγινε ε, έχουν γίνει δύο εκθέσεις σχετικές από την ε, Επιτροπή Μεταφορών. Μία από τον κύριο Πίτσεκ από τους Λέσφι Χόλσταν, ο οποίος ενώ δυστυχώς ε, έχει πεθάνει. Αλλά και οι δύο αυτές εκθέσεις είχαν γίνει με κύρια Επιτροπή, την Επιτροπή Μεταφορών. Πριν περάσω τώρα στις λεπτομέρειες, για να αναφερθώ λίγο στην διαδικασία, καθώς όλα αυτά θα γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 50 του κανονισμού, δηλαδή κατά κύριο είμαστε η κατά κύριο λόγο επιτροπή, αλλά η Επιτροπή Αλληλεία έχει έναν ιδιαίτερο α, ρόλο συμβουλευτικό θα λέγαμε. Γι' αυτό κάνουμε πρώτα απ' όλα μία πρόταση, ένα σχέδιο για τα γενικότερα α, θέματα και μετά θα ε, γνωμοδοτήσουν ε, οι συνάδελφοι γιατί μέχρι στιγμή υπήρχε κάποια αλληλεία βεβαίω εδώ πέρα στα θέματά μας οπότε συμφωνήσαμε τελικά να κάνουμε ένα σχέδιο νομίζω αυτό συμπεριλαμβάνεται από την αρχή μέχρι την παράγραφο 25 έχουμε συνοηθεί εδώ πέρα με τους συναδέλφους και έδωσα διαφορετική δομή από αυτά τα οποία είχε κάνει ο κύριος Πίτσικ δεν είναι πλέον κατά αλλά έχουμε μια συνολική αντιμετώπιση γιατί πιστεύω ότι όλοι θα μπορέσουμε να αποφεληθούμε από αυτό στο μέλλον εάν μπορέσουμε να βγάλουμε αυτά τα διαχωριστικά τύχη που υπάρχουν μεταξύ αυτών των τομέων και να κοιτάξουμε προς το μέλλον. Οπότε όλα αυτά αναφέρονται, μεταφορές, τουρισμός, αλληλεία, υπάρχει από μία παράγραφος αν θέλετε για το καθένα, αλλά όχι χωριστά κεφάλαια και όσον αφορά την ε, Επιτροπή μας είχαμε και την έκθεση Φαντάλεν για την στρατηγική των ε, θαλασσίων συγκοινωνιών για το προσχεσμένο για το 2018. Υπάρχουν αρκετά πράγματα για την ε, προστασία του κλίματος και για διάφορους άλλους τομείς. Οπότε νομίζω έχουμε αρκετές εκθέσεις στις οποίες μπορώ και εγώ να βασιστώ και αυτό είχα αυτή τη γενική προσέγγιση και επίσης για τη διαδικασία Ε, είδα το τι υπήρχε στην Γαλάζια Βίβλο, τι είχε ζητήσει το 2007 το Κοινοβούλιο, τι έχει εφαρμοστεί, τι είναι ακόμα η υποπροετοιμασία, τι υπήρχε στο πακέτο 2009 της Κομισιόν για να τα αναπτύξω όλα αυτά. Αυτές είναι οι διάφορες, από εκεί προέκυψαν διάφορες απαιτήσεις, οποίες τώρα θα αναφερθώ. Πρώτον λοιπόν, ζήτησα γιατί ακριβώς η Ευρώπη όσον αφορά την αυπήγηση πλοίων και ειδικά την πράσινη ναυτιλία και όσον αφορά τις υπεράκτητες εγκαταστάσεις έχει έναν ηγετικό ρόλο να αναπτύξει μέχρι το 2013 η Κομισιόν μια ολοκληρωμένη στρατηγική για να αναπτυχθεί αυτός ο τομέας. Το επόμενο το οποίο προέκυψε κατά τη διάρκεια της σύνταξης ήταν η καταστροφή στον κόλπο του Μεξικού και αναρωτήθηκα τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στην Ευρώπη σε μια τέτοια περίπτωση γιατί θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιδράσουμε άμεσα και να δούμε ποιοι νόμοι θα πρέπει να επανεξεταστούν για να είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι εάν συμβεί κάτι τέτοιο σε εμά. Κατόπιν ζητάω βεβαίως να διατηθούν κονδύλια για την ολοκληρωμένη θανάση πολιτική. Το ανέφερε ήδη η κυρία Επίτροπος πώς το έχει κατά νου και θα, διαθε... θα ήθελε να διαθέσει 40 εκατομμύρια για την περίοδο αυτή των δύο ετών. Κατόπιν εάν έχει νόημα να συσταθεί ένα ταμείο ακτών μια ιδέα η οποία ξεκίνησε από την Επιτροπή των Περιφερειών και εδώ πέρα εγώ ζητάω να εξεταστεί αν έχει κάποιο νόημα ένα τέτοιο ταμείο εκτών για να καλύψει όλους αυτούς τους τομείς της οικονομίας όσον αφορά τώρα την διακυβέρνηση για την πολιτική την θαλάσσια εκεί πέρα όλα τα κράτη-μέλη που έχουν ε, τέτοιες περιφέρειες και οι Κομισιόν να δουν εάν υπάρχουν τέτοιες δομές, εάν δεν υπάρχουν να τις δημιουργήσουν αλλιώς να τις εντείνουν. Επίσης θα πρέπει να ονομαστούν τα παραδείγματα που είναι οι βέλτιστες πρακτικές, οι υποδειγματικές πρακτικές που έχουν αποδειχθεί σωστές σε κάποια κρατημέλη να γνωστοποιηθούν και στα υπόλοιπα. Επίσης χρειαζόμαστε κάποια σημεία επαφής για την ολοκληρωμένη θανάσια πολιτική στα κράτη-μέλη. Κάπου υπάρχουν, κάπου δεν υπάρχουν. Ίσως θα έπρεπε να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα εκεί όπου δεν υπάρχει για ανταλλαγή ε, πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερομένων. Επίσης βεβαίως υπάρχει και αυτό το δίκτυο των ε, θαλασσίων πόλων όπου πραγματικά λειτουργούν. Εκεί πέρα συναντιούνται οι εφοπλιστές, οι αλληλείς, ε, τα ναυπηγεία, όσοι ζουν στι παράκτητε περιοχέ και εκεί πέρα θα πρέπει να αναπτύξουν την κοινή θαλασσία πολιτική. Επίση, μιλήσατε, κύριε Επίτροπε, για τι διάφορε στρατηγικέ. Στρατηγική τη Βαλτική υπάρχει, τη Βόρεια Θάλασσα συζητείτε. Οπότε πρέπει να δούμε στι περιφερειακέ στρατηγικέ όπου συζητούνται πάντα να ακολουθήσουμε και να εφαρμόσουμε αυτή την ολοκληρωμένη πολιτική γιατί για μένα είναι μια αμοιβαία υποφελής στρατηγική Στη Δε Μεσόγειο έχουμε την ιδιαίτερη περίπτωση της μεσογειακής στρατηγικής και υπάρχουν βεβαίως διαφορετικά καθεστώτα όσον αφορά την επικράτεια και την ε, κυριαρχία. Πρέπει να βρεθεί μια λύση εκεί πέρα. Αυτό μπορεί να γίνει με τη βάση την ε, σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Όσον αφορά τώρα την χωροταξία, το είπα και στην αρχή, θα πρέπει να συνοηθούμε, να δούμε ποιος τομέας της θάλασσας χρησιμοποιείται, γιατί και τι άλλο δεν μπορεί να γίνει ταυτόχρονα εκεί πέρα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια οδηγία για τη θαλάσσια χωροταξία. Ζήτησα από την Κομισιό να υποβάλει ένα σχέδιο οδηγίας μέχρι το 2011, στο οποίο θα μπορέσουν όλοι μετά να προσανατολιστούν. Κυρία Επίτροπε, μιλήσατε επίσης για το ότι οπωσδήποτε χρειαζόμαστε δεδομένα για τη θαλάσσια επιτήρηση και να δούμε βεβαίως πώς θα προστατεύσουμε και τα δεδομένα, αλλά για να ανταλλάξουμε τις πληροφορίες οποίε οποίες χρειαζόμαστε, έτσι ώστε να έχουμε προστασία των ακτών και επιτήρηση των ακτών και βεβαίως αυτό σημαίνει και περισσότερα μέσα και κονδύλια και πιθανώς μια πλατφόρμα πληροφοριών. Τέλος, πριν ε, πάω στα διάφορα, οι ε, ακτοφυλακές, ε, υπάρχει και στη Γερμανία μια συζήτηση, ήδη και στις εκθέσεις Πίτσεκ είχε αναφερθεί αυτό, πως η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει μια μελέτη σκοπιμότητας για τη συνεργασία, ίσως και τη συνένωση των διαφόρων ακτοφυλακών, κάπου βεβαίως αυτό χάθηκε, αλλά νομίζω θα πρέπει να σκεφτούμε να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί εκεί πέρα η κατάσταση. Και τέλος, στα διάφορα, στο κεφάλαιο αυτό. Θα πρέπει να δούμε πώς διάφοροι άλλοι τομείς θα μπορέσουν να ενσωματωθούν. Πρώτα απ' όλα στρατηγική για τις αλλάσιες συγκοινωνίες μέχρι το 2018, κλιματική αλλαγή, ένα πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου, γιατί αποδεδειγμένα αυτό το λένε όλα τα οικονομικά δεδομένα, διάφορα οικονομικά Ινστιτούτα που έχουν πάρα πολύ τεχνογνωσία Έχουμε ούτω ή άλλω μεγάλη παράδοση, μπορούμε να το αναπτύξουμε αυτό και να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό που υπάρχει και χρειαζόμαστε και μια στρατηγική για τον αηφόρο τουρισμό. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα για τον τουρισμό από ό,τι έγιναν με τη στρατηγική της Λισαβόνας. Η έρευνα επίσης είναι βάση για όλους τους τομείς. Είτε μιλάμε για την υπεράκτια τεχνολογία, για την ε, γαλάζια βιοτεχνολογία, για την αυπήγηση των πλοίων και τέλος το δίκτυο αυτό των δεδομένων, το τι χρειαζόμαστε θα πρέπει να είναι διεπιστημονικό και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε είδατε, πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη έκθεση, εκτεταμένη, γιατί αγγίζει πάρα πολλού τομείς, οι οποίοι όλοι τελικά επιδρούν στην οικονομική δραστηριότητά μας και νομίζω και, στι ε, μεταφορέ και στην Επιτροπή μας, δηλαδή στα θέματα μεταφορών και τουρισμού. Ευχαριστώ. Α, ξέχασα και κάτι. Ε, έχω τελειώσει την έκθεσή μου με ερωτήματα και αυτό έγινε συνειδητά γιατί θα ήθελα να δω εάν με, ε, αν θα με ακολουθήσει το Κοινοβούλιο στην άποψή μου πως είναι μια καλή προσέγγιση ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική η οποία θα έπρεπε να συνεχιστεί. Και να δούμε εάν και οι υπόλοιποι βουλευτέ και η Κομισιόν θα κινηθούν αρκετά γρήγορα για να κάνουμε αυτό το οποίο χρειάζεται. Σας ευχαριστούμε κυρία Μάισνερ. Ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαίρεται πάρα πολύ να ακούει όρου όπω διαλειτουργικότητα, ολοκληρωμένη, ενοποιημένη πολιτική. Θέλουμε απλώ να σα το πούμε αυτό. Ο κύριο Κουμουτσάκο έχει το λόγο εξ ονόματος του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου την Επίτροπο κυρία Δαμανάκη στην ε, σημερινή συνεδρία της Επιτροπής μας. Ακούσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ευαισθησία της να μην ε, εμπλέκεται όπως η ίδια είπε στο σκληρό πυρήνα των αναμειδιοτήτων των συναδέλφων της ε, κυρίων Κάλλας και Ταγιάννη αλλά απ' την άλλη εμείς και προσβλέπουμε και ενθαρρύνουμε την μεγαλύτερη επικοινωνία σας και την συνεργασία σας με την λογική ότι και οι μεταφορές και ο τουρισμός είναι δύο πολύ σημαντικά συστατικά στοιχεία της ε, ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Ε, παρά το γεγονός ότι η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της Ευρώπης είναι μια πολύ νέα ε, και σύνθετη ευρωπαϊκή πολιτική, έχει ήδη επιτύχει πρώτον να μεταβάλει τον τρόπο που σκεφτόμαστε σχετικά με τη θάλασσα, τα ζητήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε εκεί και δεύτερον έχει μεταβάλει και τον τρόπο με τον οποίο ενεργούμε όταν αναζητάμε τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Προβλήματα που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον, τη θαλάσσια οικονομία και την ασφάλεια και βεβαίως τις μεταφορές. Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική είναι μια φιλόδοξη πολιτική, αναφυσβήτητα. Γι' αυτό και εμείς, εδώ στο Κοινοβούλιο, ή μάλλον θα έλεγα πρωτίστως εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οφείλουμε να είμαστε φιλόδοξοι στους στόχους μας. Αλλά και στις προτάσεις και τις απαιτήσει μας προς την Επιτροπή αλλά και προ τα κράτη-μέλη. Και το τονίζω αυτό, ειδικά το τελευταίο, γιατί συχνά κράτη-μέλη, και δεν ξέρω τη χώρα μου, την Ελλάδα, που είναι μια κατεξοχήν θαλάσσια χώρα, πολύ συχνά λοιπόν κράτη-μέλη δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά και με τον ανάλογο ενθουσιασμό που θα έπρεπε στους στόχους που έχει θέσει η ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική. Γι' αυτό πιστεύω ότι η πρώτη προτεραιότητα που πρέπει να δώσουμε και η πρώτη προτεραιότητα της έκθεσης που συζητάμε σήμερα είναι να τονίσουμε ακριβώς αυτό το στοιχείο. Ότι πρέπει να πιεστούν και οι Επιτροπή και τα κράτη-μέλη για μεγαλύτερη ανταπόκριση. Για ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και με συγκεκριμένα βήματα εφαρμογή της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο της ανάγκης μεγαλύτερης ανταπόκρισης θα πρέπει να δούμε και ειδικότερους στόχους και επιδιώξεις. Πρώτον, θα ήθελα να αναφερθώ στην θαλάσσια διακυβέρνηση. Πρέπει να παραδεχθούμε, κυρία Επίτροπε, ότι η πρόοδο που έχει γίνει στην εφαρμογή τη δεν είναι ακόμα ικανοποιητική. Υπολείπονται σοβαρά βήματα για μια αποτελεσματική θαλάσσια διακυβέρνηση. Γι' αυτό το λόγο θα συμφωνήσω με την ε, εισηγήτρια της εκθέσεως, ε, τη συνάδελφο την κυρία Μέισερ, ότι πρέπει να γίνει μια διεξοδική αξιολόγηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των δομών θαλάσσιας διακυβέρνηση στα κράτη-μέλη, αλλά και στην Επιτροπή και στις περιφέρειες. Τα κράτη οφείλουν, ε, κυρία Επίτροπε, και εκεί η Επιτροπή έχει ένα, ένα πρόσθετο λόγο και ρόλο, τα κράτη-μέλη οφείλουν να ορίσουν το ταχύτερο δυνατό εθνικά σημεία επαφής, contact persons ή contact ε, ε, institutions, όσον αφορά την εφαρμογή της ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική αυτή η ολιγορία πολλών κρατών μελών να προχωρήσουν σε δομές θαλάσσιας διακυβέρνησης είναι ενοχλητική και εν μέρει ακατανόητη. Όσον αφορά τις περιοχές και τις θαλάσσιες λεκάνες, είναι σαφές ότι ειδικότερη προσοχή πρέπει να δώσουμε στη Μεσόγειο. Γνωρίζουμε όλοι τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, την οικονομική, την τουριστική και πολιτιστική της και πολιτική της σημασία. Αρκεί μόνο να φέρει κανείς έναν αριθμό, το 30% του παγκοσμίου εμπορίου που γίνεται δια θαλάσσης συγκεντρώνεται στην Μεσόγειο. Όμως, έχουμε ένα πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε για μια εφαρμογή πρακτικών πολιτικών στη Μεσόγειο. Και αυτό το πρόβλημα είναι ότι λόγω της μη υπογραφής και μη κύρωσης και επομένως της μη εφαρμογής της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας από όλα τα παράκτια κράτη, ορισμένα εκ των οποίων μάλιστα ε, διεκδικούν και έχουν και σχέσεις στενές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάω και για υποψήφια κράτη, δεν έχουν προχωρήσει σε αυτή την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας. Και αυτό είναι σοβαρή τροχοπέδη. Είναι σοβαρή τροχοπέδη διότι δεν έχουν προκύψει οι ανιαγκαίες οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και έτσι μεγάλο τμήμα της Μεσογείου είναι ουσιαστικά ένα no man's land και επομένως εκεί πέρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί καμία συγκεκριμένη πολιτική στο πλαίσιο της λογικής της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ευρώπης. Θαλάσσια επιτήρηση. Η Επιτροπή θα πρέπει, όπως άκουσα και είναι στο στόχο σας, να παρουσιάσετε έναν οδικό χάρτη για την εφαρμογή της από τα κράτη-μέλη. Αλλά ίσως αυτό να μην είναι αρκετό. Πρέπει να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά και θα πρέπει να ξεκινήσει η Επιτροπή να δουλεύει για τη διαμόρφωση ενός νομικού πλαισίου που θα επιτρέπει την ενοποίηση τη θαλάσσια επιτήρηση. Πώ θα αλλάζουμε στοιχεία, γιατί υπάρχουν ορισμένα νομικά θέματα που προκύπτουν, ειδικά όσον αφορά την ανταλλαγή ε, στοιχείων και ολοκληρωμένη ενημέρωση. Κλείνω, κυρία Επίτροπε, με ορισμένε ε, παρατηρήσει για την έκθεση τη συναδέλφου τη κυρία Μέισερ. Υπάρχουν σημεία στα οποία θα θέλαμε να είναι πιο φιλόδοξη η έκθεση αυτή. Θα θέλαμε, παραδείγματο χάρη, να υπάρχει μια πληρέστερη αναφορά στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό. Είναι σημαντικό ότι με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε πια τη νομική βάση για μια ευρωπαϊκή πολιτική τουρισμού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας και να το αξιοποιήσουμε. Και να εντάξουμε στην έκθεση αυτή πληρέστερες αναφορές και πιο συγκεκριμένες αν είναι δυνατόν κατευθύνσεις για τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό. Θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα, επίσης σημαντικός τομέας. Ο τομέας ενέργειας, στη θάλασσα. Είναι πολύ σημαντικό. Και ειδικά για τι βιώσιμε και εναλλακτικέ πηγέ ενέργεια. Θα μιλήσω εδώ ειδικά, θα αναφερθώ εδώ ειδικά στην αιωλική ενέργεια στη θάλασσα. Είναι μια πολύ σημαντική, ένας πολύ σημαντικός τομέας ε, που επίσης θα πρέπει να δούμε. Μιλώντας για εναλλακτικέ πηγές ενέργειας, άρα φιλικές στο περιβάλλον, δεν μπορώ παρά μην αναφερθώ ιδιαίτερα στο μεγάλο ατύχημα δυστύχημα στον κόλπο του Μεξικού. Κύριε Επίτροπε, είναι βέβαιο ότι οι αμερικανικές αρμόδιες αρχές και η κυβέρνηση έχει καταλήξει σε ορισμένα συμπεράσματα από τη διαχείριση της κρίσης. Υπάρχουν ορισμένα lessons learned. Πιστεύω ότι αυτά θα πρέπει να τα δούμε κι εμείς και ενδεχομένως να τα αξιοποιήσουμε προσαρμοζόντας τα βέβαια στις δικές μας συνθήκες και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Γι' αυτό, κυρία Επίτροπη, ίσω θα ήταν μια χρήσιμη ιδέα, την οποία μπορείτε να αξιολογήσετε και μαζί με του συναδέλφου σα επιτρόπου, να γίνει μια επαφή με τι Αμερικανικέ Αρχέ από πλευρά Επιτροπή. Να μα ενημερώσουν ποια ήταν τα προβλήματα, ποιε ήταν ε, οι αδυναμίε και ποια ήταν ε, τα μέτρα εκείνα που θα έπρεπε να έχουν ληφθεί εγκαίρω ώστε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τέτοιου είδου ε, πολύ δυσχερεί και ανησυχητικέ καταστάσει. Βεβαίως ε, ε, από πλευρά ναυτιλία υπάρχουν τα πακέτα έρικα και η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει πολλά σοβαρά βήματα. Αλλά δεν επαρκεί αυτό. Κλείνω κύριε Πρόεδρε, βλέπω το, ότι κουνάτε το σφυρί τη λήξη του χρόνου, αλλά θα μου δώσετε δύο λεπτά ακόμα, ελπίζω στην κατανόησή σα. δημοσιονομικε προοπτικες προοπτικές 2013-2020. Πρέπει να εντάξουμε τη στρατηγική, τη θαλάσσια με φιλοδοξία εκεί, ειδικά για νησιωτικέ περιοχέ και για το Ταμείο Ακτών. Κύριε Πρόεδρε, πήρα λίγο περισσότερο χρόνο γιατί οι Έλληνε έχουμε μια ευαισθησία για τη θάλασσα. Άλλωστε χρησιμοποιούμε την ίδια λέξη θάλασσα, απαράλλακτη με τα ίδια γράμματα και την ίδια προφορά 3.000 χρόνια τώρα. Γι' αυτό και αυτή η ευαισθησία κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την κατανόησή σα. Η κυρία Τικάου για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια καθώς επίσης και την Επίτροπο για την παρουσία της εδώ σήμερα. Θα ήθελα να μιλήσω εξ ονόματος του συναδέλφου μου του κυρίου Κνούτ Φέκενστάιν, ο οποίος δεν μπορεί να είναι παρόν σήμερα και είναι ο σκιώδης συγητής εξ ονόματος των σοσιαλιστών. Θα μιλήσω στα αγγλικά προκειμένου να είμαι όσο δυνατόν πιο ακριβής για να σας πω ουσιαστικά αυτά που θα ήθελα να σας πει ο κύριος Κνούτε. Αγαπητοί ε, συνάδελφοι, αγαπητοί συγγήτρια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκθεση αυτή σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Η ομάδα των ε, σοσιαλιστών και δημοκρατών είναι υπέρ της πολιτικής αυτής, όπως άλλωστε και η συγγήτρια. Και όπως είπε και η συγγήτρια, πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στο ζήτημα της διακυβέρνησης και της διοικητικής δομής και ότι ε, θα πρέπει στους επιμέρους τομείς να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα μέτρα τα οποία αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εφαρμόζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τον καλύτερο δυνατό συντονισμό. Όσον αφορά την ε, στρατηγική τη θαλάσσια για το 2018, πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιμέρους λεπτομέρειες, επομένω όντως θα πρέπει να έχουμε μια στονισμένη προσέγγιση. Ωστόσο θα ήθελα να σας πω κάτι το οποίο συνδέει την ε, διακυβέρνηση και τις κυβερνητικές δομές με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Αν δούμε την καταστροφή με την πετρελοκυλίδα στι ΗΠΑ μου δημιουργούνται πάρα πολλέ ανησυχίε. Η κυρία Μάισνερ στο άρθρο 4 λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αντλήσει τα απαραίτητα διδάγματα από την καταστροφή αυτή λόγω της πετρελοκυλίδας. Η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών συμφωνεί με αυτό και όντως χρειάζονται περισσότερες διευκρινήσεις για το ζήτημα αυτό και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση. Από την πλευρά λοιπόν των σοσιαλιστών θα θέλαμε να συμπεριληφθεί το άρθρο αυτό. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχει συμπεριληφθεί μάλλον, αλλά χρειάζεται επίσης και μία λεπτομερής ανάλυση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς έχουν σήμερα τα πράγματα στην Ευρώπη. Προβλέπετε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης αν κάτι τέτοιο συμβεί και στην Ευρώπη. Είναι τα δηληστήρια offshore της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασφαλή. Υπάρχουν νομοθετικά κενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία θα πρέπει κατεπηγόντως να καλύψουμε. Αυτά τα σημεία λοιπόν θα πρέπει να εξετάσουμε και επίσης στα πλαίσια της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής θα πρέπει να διευθετηθούν και αυτά. Επίσης θα ήθελα να αφαιρθώ και στο άρθρο 28 όπου αναφερόμαστε εδώ πέρα στο πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε καλύτερη ασφάλεια, καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, καλύτερη προστασία του τομέα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε την εξέλιξη της ΕΜΣΑ στα πλαίσια της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Νομίζω ότι ακόμα υπάρχουν κάποιες δυνατότητες, κάποιες ευκαιρίες όπου θα μπορούσαμε να εμπλέξουμε την ΕΜΣΑ με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεση αυτή. Η ψηφοφορία από ό,τι βλέπω θα γίνει το Σεπτέμβριο, επομένως έχουμε ακόμα κάποιο χρόνο μπροστά μας για να εργαστούμε από κοινού. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία ο κύριος Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, και καλώς ήρθατε με την αρμοδιότητά σας σε όλους αυτούς τους τομείς. Όταν ε, ε, ήσασταν υποψήφια για τη θέση της Επιτρόπου, Είχαμε κάποιες επιφυλάξεις ε, για το κατά πόσο ήσασταν αρμόδια να καταλάβετε αυτή τη θέση. Δεν, ήμουν καθόλου, ε, δεν ήμασταν καθόλου σίγουροι κατά πόσο θα μπορούσατε να επιληφθείτε αυτού του νέα. Τώρα όμως που είσαστε η νέα Επίτροπος Θαλάσσιων Μεταφορών ε, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ίσως υπάρχει μια μικρή σύγκρουση συμφερόντων με τον κύριο Κάλλας. αλλά ας ελπίσουμε να μην υπάρχει και σύγκρουση αρμοδιοτήτων με τον τομέα του κύριου Τατζάνη στον τουρισμό. Ε, ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων μοιάζει να είναι αρκετά περίπλοκος και για πρώτη φορά βλέπουμε κάτι τέτοιο στην έκθεση της κυρίας Μάισνερ. Φαίνεται να επικρατεί μεγάλη σύγχυση σε αυτό το διάβημα της ολοκλήρωσης η Επιτροπή μας θα πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα των θαλάσσιων μεταφορών και φυσικά η έκθεση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά απλώνεται σε πολλά και διαφορετικά ζητήματα. Το ζήτημα λοιπόν είναι εμπίπτουν όλα αυτά στον τομέα των, δραστη... των αρμοδιοτήτων μας στο πεδίο των αρμοδιοτήτων μας. Μήπως ε, έχουμε βγει έξω από τα όρια των αρμοδιοτήτων των ε, αρμοδιοτήτων μας. Ο κόσμος μας είναι πάρα πολύ ακριβός. Η... Αν η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική πρέπει να καλύψει όλους αυτούς τους διαφορετικούς τομείς, ε, η, η, η συγγήτρια ζητά τη γνώμη μας. Εάν η ολοκληρωμένη λοιπόν θαλάσσια πολιτική πρόκειται να καλύψει όλους αυτούς τους διαφορετικούς τομείς, θα πρέπει να επεκταθούμε και να μιλήσουμε και για τα ναυπηγεία, όπου έχει μειωθεί η δραστηριότητα κατά 80%. Πρέπει να μιλήσουμε για την θαλάσσια ρήπανση, όχι μόνο για στον κόλπο του Μεξικού, αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να επισέλθουμε στην Μεσόγειο όλος ιδιαιτέρως. Αναρωτιέμαι όμως εάν οι φιλοδοξίες μας εναρμονίζονται με, την, με τους κανόνες που διέπουν ε, το αντικείμενό μας, το πεδίο των αρμοδιοτήτων μας. Και με βάση την έκθεση της κυρίας Μάισνερ θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για πολύ περισσότερα πράγματα ακόμη προετοιμαζόμαστε, ε, προετοιμάζουμε κάποιες τροπολογίες πολύ καλόπιστα για να βελτιώσουμε αυτή την πάρα πολύ καλή έκθεση. Just... Ε, πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, βλέπω κάποια ονόματα αγοριτών που θέλουν να, λάβουν και πάλι το δεύτερο, που θέλουν να δευτερολογήσουν. Αν έχουμε χρόνο θα τους επιτρέψουμε να δευτερολογήσουν Πρώτα όμως θα εξαντλήσουμε τον κατάλογο των αγοριτών που έχουν ζητήσει πρώτη το λόγο. Λοιπόν, όποιοι θέλουν να δευτερολογήσουν θα τους γράψω στο κάτω-κάτω μέρος του καταλόγου. Κύριε Ντανέλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω την Επίτροπο, την κυρία Δαμανάκη, ε, για τη συνεργασία της με την Επιτροπή μας. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει εξάλλου ότι η κυρία Δαμανάκη κατάγεται από μια νησιωτική περιοχή, από την Κρήτη. Έτσι έχει βιωματική σχέση με τα προβλήματα που η ένταση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων δημιουργεί στις παράκτες ή στις θαλάσσιες περιοχές και άρα αντιλαμβάνεται απολύτω και την αναγκαιότητα της υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Οι δράσεις που προωθούνται στο πλαίσιο της ε, ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής αξιοποιούν σημαντικές συνέργειες που προκύπτουν από το φάσμα των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, όσο και αν αυτές ε, διαπλέκονται μεταξύ τους και κάποιες ίσως είναι και, ε, έχουν και αντιφατικά αποτελέσματα στην εξέλιξή τους. Νομίζω ότι η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική μας δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε σάρκα και οστά και στο στόχο της μπλε ανάπτυξης, διαμορφώνοντας μηχανισμού συντονισμού των αναγκών της αλληλεία, των μεταφορών, της έρευνας του τουρισμού, προωθώντας τη συγκρότηση κοινών στοιχείων και γνώσεων μεταξύ των επιμέρους τομέων και βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες μεταξύ των περιφερειακών θαλασσών όπως είναι η Βαλτική ή η Μεσόγειος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στήριξε εξ αρχής τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και πιστεύω θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υλοποίησής της να αναφερθώ ότι θεωρώ ιδιαίτερη σημασία έργα για την επιτυχή έκβαση της ε, ολοκληρωμένης θαλάσσης πολιτικής αποτελούν τα διατομεακά οριζόντια εργαλεία που βρίσκονται υπό διαμόρφωση, κυρίως ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, στον οποίο αναφέρθηκε και η Επίτροπος, θα πρέπει να μας επιτρέψει να διαχειριστούμε με ισόρροπο τρόπο τις ολοένα και πιο εντατικές χρήσεις θάλασσας, δεδομένη ειδικά και τη αυξανόμενη άντληση των ανανέσιμων πηγών ενέργεια από θαλάσσιε παράκτιε περιοχέ, είτε από τον κυματισμό είτε την αιωλική, να συνδυάσουμε την ανάπτυξη στου επιμέρου τομεί με τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεών του, που είναι και το σημαντικότερο ε, πρόβλημα τη ανάπτυξη των όποιων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον και να εισάγουμε στα παραπάνω ένα διασυνοριακό και διαπεριφερειακό συντονισμό που σχεδόν ολοκληρωτικά πουσιάζει μέχρι σήμερα. Τα μέτρα που φέρνει η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, αλλά και οι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ πολιτικέ για τη θάλασσα, μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα τη μπλε ανάπτυξη, φτάνει να οθήσουν κυβερνήσει, περιφέρειε και επιχειρήσει να αγκαλιάσουν τη διασυνοριακή και διατομεακή θαλάσσια συνεργασία. Κλείνοντα, θα ήθελα να ρωτήσω την Επίτροπο πώς η Επιτροπή βλέπει να ενισχύεται η θαλάσσια διακυβέρνηση με την ουσιαστική και μόνιμη ένταξη ε, στις δομές της ε, θαλάσσιας διακυβέρνησης όλων των εμπλεκομένων, δεδομένης της, ε, όπως βλέπουμε, ολιγορίας των εθνικών αρχών στην συμμετοχή τους σε μία αντίστοιχη κοινή προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Δανέλη. Κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την κυρία Επίτροπο, την κυρία Δαμανάκη για τις εξηγήσεις μας έδωσε. Ευχαριστούμε και την κυρία Μάισνερ για την ε, έκθεσή της. Σε γενικές γραμμές ε, πράγματι πρέπει να είναι ολοκληρωμένη η θαλάσσια πολιτική. Μιλάμε για τις μεταφορές, το περιβάλλον, την αλληλεία, την ενέργεια, τη βιομηχανία και από ό,τι φαίνεται όλα αυτά σε τελική ανάλυση είναι αλληλένδετα και συμφωνώ με μία από τις πτυχές στην οποία αναφέρατε η οποία είναι η καινοτομία γιατί πραγματικά εάν μιλάμε για κάτι σε αυτή την οικονομική κρίση και την στρατηγική του 2020 είναι πραγματικά πως ε, πρέπει να τονίσουμε το θέμα της ε, καινοτομίας. Η καινοτομία στον τομέα των θαλάσσιων είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε με κανένα τρόπο. Έχω όμως ε, μια ερώτηση και ένα σχόλιο και μια αξιολόγηση που θα ήθελα για τα εξής. Πρώτα απ' όλα, είμαστε ή δεν είμαστε σε θέση να εγκρίνουμε ένα έγγραφο το οποίο μιλάει για ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, το οποίο θα είναι χρήσιμο δεν έχω μεγάλη εμπειρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι εδώ πέρα λιγότερο από ε, τόσο, αλλά αυτό το οποίο βρίσκω εντυπωσιακό είναι ότι εγκρίνουμε πάρα πολλά έγγραφα με ερωτήσεις, αλλά σπάνια μπορούμε πραγματικά να αποφασίσουμε σε, για πράγματα τα οποία είναι τόσο συγκεκριμένα ώστε να μπορούν να δουν αυτά αποτελέσματα οι Ευρωπαίοι πολίτες αν το συνδυάσουμε αυτό και με την κρίση και με τη στρατηγική του 2020, νομίζω θα πρέπει να φροντίσουμε αυτά τα μέτρα να είναι πιο άμεσα όσον αφορά τα αποτελέσματα. Τώρα, μιλήσατε για την ανάγκη μιας μελέτης για να δούμε ποιες είναι οι νέες ευκαιρίες για τις ε, θέσεις εργασίας, για δουλειές οι οποίες ε, είναι και παραδοσιακές ε, εάν θέλετε και δεν έχουν αλλάξει όπως στον τομέα της αλληλείας και της βιομηχανίας και βλέπουμε πως υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι καινοτόμε και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και νέου είδους ε, θέσεις εργασίας ε, και αυτά κυμαίνονται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι την έρευνα για νέα προϊόντα και τη βιοτεχνολογία. Μιλά, μιλήσατε επίσης για το 2012 όσον αφορά τη σύνταξη αυτής της έκθεσης. Οι παράκτιες περιοχές οι οποίες προχωράνε ήδη σε αυτά τα έργα ε, θα ενταχθούν σε αυτή την ε, πολιτική, θα φαίνονται σε αυτή την πολιτική που συντάσσουν ήδη οι υπηρεσίες σας π.χ. συγκεκριμένα για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους χωρίς να περιμένουμε το 2012 και ένα ακόμα ερώτημα είναι ποιο είναι το μέλλον ε, και ποια η προσέγγιση που θα ακολουθήσει η Κομισιόν θα θέλαμε να μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε σε ένα έγγραφο. Θα ήθελα λοιπόν να να σας ρωτήσω για το έγγραφο αυτό της ολοκληρωμένης πολιτικής. Αυτό είναι ένα έγγραφο το, στο οποίο έχουν συμφωνήσει και οι υπηρεσίε τουρισμού, μεταφορών ε, κτλ. Γιατί μιλάμε όντως για ολοκληρωμένη πολιτική, οπότε πρέπει να συμφωνήσουν και οι άλλες υπηρεσίες και αυτό βεβαίως σημαίνει πως πρέπει να εμπλακούν και οι περιφέρειες γιατί αυτές αφορά η ευρωπαϊκή πολιτική, αν δεν μπορέσουμε να σωματώσουμε τις περιφέρειες στην ευρωπαϊκή πολιτική, να τα φέρουμε όλα αυτά στο τοπικό επίπεδο, τότε δεν λαμβάνουμε τις σωστές αποφάσεις και δεν διαχειριζόμαστε τα πράγματα αποτελεσματικά. Πολλές ε, περιφέρειες έχουν προχωρήσει πέρα από τα κράτη-μέλη σε αυτό τον τομέα. Και αυτό σχετίζεται με την ανταλλαγή πληροφοριών και τις βελτιστές πρακτικές. Δεν χρειάζεται να εφεύρουμε ξανά τον τροχό εδώ πέρα. Χρειάζεται λίγη καινοτομία στην Ευρώπη. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε διαφορετικά ασφάλειας και από ατυχήματα και από κακόβουλες ενέργειες. Το αναφέρατε και πιο πριν. Στο έγγραφο αυτό, στην ολοκληρωμένη αυτή πολιτική, δεν έχω δει τίποτα για το ζήτημα της ασφάλειας, που είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αποτελέσει τμήμα της πολιτικής αυτής. Έχουμε πλοία που ψαρεύουν σε ύδατα τρίτων χωρών, πλοία που απολαμβάνουν ειδική προστασία και αυτό σημαίνει πως επηρεάζονται εδώ πέρα και άλλοι τομεί. Οπότε αν μπορούμε να έχουμε ασφάλεια για τα ληφτικά αυτά σκάφη, εδώ πέρα νομίζω θα ήταν κάτι το πολύ χρήσιμο. Τώρα, εμείς είμαστε υπέρ στους ολοκληρωμένες πολιτικής, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε ενισχυμένο συντονισμό μεταξύ μας και εντός της Κομισιόν πρέπει να το κάνετε αυτό και να είναι σαφές ότι η Κομισιόν συμφωνεί στο τι σημαίνει η ολοκληρωμένη θανάσια πολιτική έτσι ώστε να μπορέσει και το Κοινοβούλιο να δουλέψει πιο εντατικά στις διάφορες επιτροπές. Πρέπει να γνωρίζουμε ποιο είναι πραγματικά το, ο ευρωπαϊκός στόχος εδώ πέρα. Αλλιώ, σύμφωνα με τη σύντομη βεβαίως εμπειρία μου, θα συνεχίσουμε να το συζητάμε αυτό μεταξύ των διαφόρων ομάδων και κρατών μελών, αλλά δεν θα προκύψει τίποτα και δεν μας περισσεύει χρόνος, οπότε θα πρέπει να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια να έχουμε ένα έγγραφο το οποίο θα μπορέσει να αποτελέσει ένα υπόδειγμα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Νομίζω πως ε, στον τομέα αυτό πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο ευρωπαϊκό μοντέλο αντί να δημιουργούμε περαιτέρω συγκρούσεις μεταξύ ομάδων ή και ε, επιτρόπων. Σας ευχαριστώ, κύριε Στέιλορ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Κυρίε και κύριοι, είναι η πρώτη συνεδρίαση στην οποία λαμβάνω μέρος, οπότε δεν είστε μόνο εσείς οι νέα πλέον, είμαι και εγώ καινούριο. Είμαι βουλευτής εδώ και τρεις εβδομάδες και βεβαίως ε, ελπίζω να συνεισφέρω και εξ ονόμου των Πρασίνων καλωσορίζει τη γενική κατεύθυνση της έκθεσης την οποία υποστηρίζουμε. Καλωσορίζουμε ιδιαίτερα το ότι αναφέρεται η ενσωμάτωση διαφόρων υπηρεσιών άκτοφυλακής και συγκεκριμένα στην παράγραφο 14 αναφέρονται συγκεκριμένες στρατηγικές οι οποίες θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες των θαλασσίων λεκανών. Αυτό είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζετε και νομίζω πως και η Επιτροπής κυρία Δαμανάκη το τόνισε αυτό. Έχω όμως κάποιες προτάσεις που ελπίζουμε ότι θα κάνουν την έκθεση έτσι πιο εύρωστη η ανηφορία νομίζω εδώ πέρα είναι το κοινό νήμα που διατρέχει τα διάφορα στοιχεία της ολοκληρωμένης ε, θαλάσσιας πολιτικής. Πρώτα απ' όλα λοιπόν για την παράγραφο 4 που αναφέρει την πετρελαιοκυλίδα στον κόλπο του Μεξικού εμείς θα θέλαμε να δούμε πιο έντονη διατύπωση. Π.χ. καλεί την Κομισιόν να δει όλα τα πιθανά νομοθετικά παραθυράκια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών για να προληφθεί μια τέτοια καταστροφή. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν το τι σκοπεύει να κάνει για την ασφάλεια των εξεδρών αυτών άντλησης ε, πετρελαίου, αν προγραμματίζει κάποια νομοθεσία και αν ναι πότε σκοπεύει να τη δημοσιεύσει. Επίσης, ε, για την ανάγκη αυτή αποτελεσματικής ε, προστασίας. Οι παράγραφοι 18 και 19 πρέπει να συμπληρωθούν με την αναγνώριση της ανάγκης για να δούμε ποιες είναι οι ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές, οι οποίες θα πρέπει να τύχουν ειδική προστασίας και επιτήρησης και τα πλοία με επικίνδυνα φορτία θα πρέπει να απαγορεύεται να διέλθουν από εκεί. Ταυτόχρονα, στην παράγραφο 27, θέλουμε πιο έντονο ρόλο στην προστασία του κλίματος με το να συμπεριληφθούν οι θαλάσσιες μεταφορές στο σύστημα εμπορίας εκπομπών και στους στόχους της Ευρώπης 2020. Επιπλέον, προτείνουμε η παράγραφος 17 να δώσει περισσότερο βάρος στην ε, δημιουργία και χρήση ΑΠΕ. Και εδώ πέρα εννοούμε ηλιακή, αιωλική και κυματισμού. Και αυτό και για την ε, κίνηση και για την δημιουργία ενέργειας στα πλοία. Επίσης ε, αυτό και για τις απαιτήσεις της παραγράφου 30. Οπότε τέλος χαιρόμαστε για το ότι γίνεται αναφορά στην παράγραφο 29 στον αηφόρο τουρισμό. Θα θέλαμε όμως να συνδεθεί αυτό με την αρχή της προστασίας της φύσης των παράκτιων περιοχών. Και αυτό σας το λέω εγώ που έχω ζήσει όλη μου την περιοχή σε παράκτια περιοχή στην Αγγλική ακτή. Αυτά λοιπόν και αυτή ήταν η πρώτη μου παρέμβαση. Σας ευχαριστούμε κύριε Τέιλορ. Γνωρίζουμε πως είναι πολύ περήφανοι οι Άγγλοι για τις παρθενικές τους παρεμβάσεις ε, συγχαρητήρια λοιπόν για την πρώτη σας ε, παρέμβαση. Είναι κάτι το οποίο δεν αντιλαμβάνονται οι συνάδελφοι, αλλά εγώ καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι ως Βρετανός βουλευτής. Τα συγχαρητήρια μου λοιπόν. Κύριος Κάτσιαν κατόπιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε εγώ σημείωσα και θέλω να αναφέρω δύο πραγματάκια πάνω στα οποία έχω πολλές αμφιβολίες. Εσείς, κυρία Επίτροπε, αναφέρατε στοιχεία και ημερομηνίες το 2012, το 2011 νομίζω ότι είναι πολύ μακρές αυτές, είναι πολύ μακριά αυτές οι προθεσμίες αν θέλουμε να επιτύχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Μιλήσατε για ανάπτυξη, για ανάπτυξη στο πλαίσιο της θαλάσσιας πολιτικής. Όπως είπε και η συνάδελφος Μάισνερ, ο τομέας αντιπροσωπεύει το 50% του ακαθάριστου προϊόντος. Αυτή η ανάπτυξη την οποία την εντάσσετε στο πρόγραμμά σας, πώς θα επιτύχετε επιτευχθεί αυτή η ανάπτυξη. Αναφέρθηκε ένα ταμείο για τις ακτές από την κυρία Μάισνερ. Είναι μια ιδέα να υπάρξει ένα συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο για να μπορέσουμε να συντονίσουμε κάτι σημαντικό από οικονομική άποψη. Ε, περνούμε μια δύσκολη φάση για την απασχόληση και την οικονομία. Σήμερα λοιπόν, τόσο όσο αφορά το χρονοδιάγραμμα, όσο αφορά και τις πρωτοβουλίες, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή και το σημείο χρόνος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πολλά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί για τις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές και με τα ζητήματα της αλληλείας και όσα έχουν αποφασιστεί να εφαρμοστούν από την 1η Ιουλίου και μετά. Σε αυτή τη στρατηγική λοιπόν, την προγραμματική στρατηγική, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τον χρόνο και θα ήθελα να μας πείτε κάτι παραπάνω γι' αυτό. Ευχαριστώ. Τι ήταν αυτό. Η κυρία Γιάλα Σέντερ, σα ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την παρουσίαση που έκανε και να ευχαριστήσω την κυρία Μάισνερ για την έκθεσή τη. Όσον αφορά τι κοινωνικέ πτυχέ, Θεωρώ ότι ε, ο τομέας αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός όσον αφορά την ορατότητα που έχουμε απέναντι στους πολίτες μας. Φτάνουμε στην ολοκλήρωση μιας πρώτης δέσμης μέτρων για τα δικαιώματα των ε, επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές με πολύ καλή συνεργασία και με τα άλλα δύο θεσμικά όργανα. Αυτή η πρώτη δέσμη είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει ένα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Ιδίως ε, όσον αφορά τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για τους επιβάτες, τους κατάλληλους τερματικούς σταθμούς θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ή θα μπορούσαμε να προσαρμόσουμε τους υφιστάμενους. Στον τομέα της θαλάσσιας πολιτικής γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά επαγγελματικά προβλήματα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα εξυγχρονισμού και δεν καταφέρουμε να προσελκύσουμε αρκετούς νέους. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω τι προτίθεστε εσείς να κάνετε. Σαφώς μπορεί κάτι να γίνεται για τους καπετάνιους ή για τους πιλότους, αλλά αυτοί αν θέλετε αποτελούν λίγο την αφρόκρεμα. Τι θα γίνει για τους υπόλοιπους που βρίσκονται στις άλλες βαθμίδες των επαγγελματικών αυτών κλάδων. Επίσης, οι άκρος απομακρυσμένες περιοχές στην Ευρώπη. Αυτές διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στα πλαίσια της θαλάσσιας πολιτικής, μόνο ότι απέχουν πάρα πολύ από το κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα λοιπόν να γνωρίζω τι θα κάνετε για αυτές τις ε, περιοχές που βρίσκονται ιδιαίτερα μακριά, τις άκρο απότερε περιοχές. Επίσης, θα θέλαμε να δούμε ποια είναι η έρευνα η οποία θα μπορούσε να γίνει στον ε, πυθμένα των θαλασσών, έρευνες που θα μπορούσαν να γίνουν ε, έρευνες θα μπορούσαν να γίνουν και σε ναυάγια. Επίσης, ε, πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αρχίσει να επεξεργαζόμαστε τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές και θα θέλαμε η θαλάσσια πολιτική να έχει ένα μεγαλύτερο τμήμα πλέον του κοινοτικού προπολογισμού. Αυτό Αποτελεί αρμοδιότητα λοιπόν τη Επιτρόπου και θα θέλαμε εμεί να γνωρίζουμε πώ θα μπορούσαμε να σα βοηθήσουμε προκειμένου να αυξηθεί ο κοινοτικό προπολογισμό για τη θαλάσσια πολιτική. Δεν θέλουμε συνολική αύξηση του προπολογισμού, αλλά θέλουμε ένα μεγαλύτερο μερίδιο του υφιστάμενου προπολογισμού να δίνεται στη θαλάσσια πολιτική. Η κυρία Τικάου πάλι έχει το λόγο, θα μιλήσει αυτή τη φορά εκπροσωπώντα τον εαυτό τη και όχι τον κύριο Φλέκενστάιν. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Θα ήθελα να πω ότι το χρονοδιάγραμμα το οποίο ανέφερε η κυρία Μάισνερ στο άρθρο 3 ζητά ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τα τέλη του 2013 να παρουσιάσει μια στρατηγική διατομεακή για τις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές. Θεωρώ ότι το έτος 2013 είναι πολύ μακριά. Νομίζω ότι η στρατηγική αυτή θα πρέπει να προταθεί το αργότερο στα μέσα του 2011. Και αυτό γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημιούργησε μία επιτροπή για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές και εντολή αυτής της νέας επιτροπής θα ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2010 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2011. Στόχος της νέας αυτής επιτροπής είναι να τεθούν οι σωστές βάσεις για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον ένα σχέδιο, ένα προσχέδιο της νέας αυτής στρατηγικής ε, μέχρι τα μέσα του 2011, προκειμένου να μπορούμε να τις περιλάβουμε στις νέες δημοσιονομικές προοπτικές. Θα μπορούσαμε επίσης να μιλήσουμε για τη χρήση των διευθυντικών ταμείων, είτε για τον τουρισμό, είτε για την περιφερειακή ανάπτυξη. Και έχουμε και το άρθρο 23 της κυρίας Μάισνερ, το οποίο θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμο προς αυτό. Θα ήθελα επίσης να σας πω, να κάνω μια έκκληση ουσιαστικά. θα υπάρχει κάποιο σχέδιο για την υποθαλάσσια μεταφορά υδρογοναθράκων. Κύριε Κουμουτσάκο, μιλήσατε πριν και ζητήσατε να δευτερολογήσετε. Επειδή έχουμε λίγο χρόνο, Βεβαίω, αλλά με όλο το σεβασμό ελπίζω να μην είναι η δεύτερη σα παρέμβαση τόσο μακροσκελή όσο η πρώτη. Λοιπόν, έχετε το λόγο cannot be repeated, German. Um, Ξέρετε ότι δεν επαναλαμβάνονται τα, τα πρωτότυπα. Λοιπόν, ζήτησα το λόγο για να πω πως η πρόθεσή μα εδώ πέρα είναι να υποστηρίξουμε την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, η οποία ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια και να μην ε, αρχίσουμε να αμφισβητούμε μια ολόκληρη πολιτική η οποία είναι ολοκληρωμένη. Αυτά. Ε, ήμουν αρκετά γρήγορος. Ήσασταν εξαιρετικός και σας ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Δεν θα ζητήσω να επανέλθω. Ωραία. Γιατί δεν θα σας έδινε και το λόγο. Κυρία Επιτροπέ, να προσθέσω κι εγώ λίγα λόγια. Νομίζω πως όλοι υποστηρίζουν την προσέγγιση αυτή της ολοκληρωμένης πολιτικής και όπως είπε και ο κύριος Κουμουτσάκος δεν είναι κάτι το καινούριο όσον αφορά την Επιτροπή μας και επαναλαμβάνουμε κατά κάποιον τρόπο πράγματα τα οποία έχουν ήδη υποθεί, όπως είπε και η συγκήτρια, ο κύριος Πίτσικ ε, ε, είχε κάνει τις εκθέσεις Πίτσικ 1 και Πίτσικ 2, σαν το Ράμπο. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα. Εάν ακολουθήσουμε αυτή την ε, προσέγγιση για την ολοκληρωμένη θανάσια πολιτική, για το ποιος είναι υπεύθυνο εντός του Κοινοβουλίου, και η κυρία Μάισνερ αναφέρθηκε ε, κάπως διπλωματικά στο ζήτημα που είχαμε με την Επιτροπή Αλληλείας όσον αφορά την αρμοδιότητα νομίζω πως είναι σωστό ως πρόεδρος της Επιτροπής εγώ να διεκδικήσω και τα δικά μας δικαιώματα και να πω πως όσον αφορά την Επιτροπή Μεταφορών η θαλάσσια πολιτική είναι αρμοδιότητα της ε, Επιτροπής μας. Ότι είναι κάτω από τη θάλασσα ή αντλείται από τη θάλασσα μπορεί να είναι αρμοδιότητα άλλων επιτροπών. Και το λέω αυτό γιατί γνωρίζω πως ε, η καταστροφή με την πετρελαιοκυλίδα στον κόλπο του Μεξικού είναι ένα ε, γεγονός που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στα ΜΜΕ. Και έχοντας διεκδικήσει την θαλάσσια πολιτική εξ ονόματος της Επιτροπής μας, πρέπει να υπενθυμίσω βεβαίως στους συναδέλφους μας πως είπε εξέδρες άντλησης πετρελαίου δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Είναι αρμοδιότητα άλλης Επιτροπής, Επιτροπής Βιομηχανίας. Όπως είναι και τα ναυπηγεία και τα διαλυτήρια πλοίων, τα οποία είναι όντω και αυτά αρμοδιότητα τη Επιτροπή Βιομηχανία και βεβαίω οι ναυτικοί οι συνθήκες εργασίας κτλ. Αυτά είναι θέματα τη επιτροπή απασχόληση. Οπότε από την φύση της ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική κάτι το οποίο θέλουμε, Ήδη αυτομάτω πρέπει να διευρύνουμε και την δική μας έντολη, να συμπεριλάβουμε και άλλε επιτροπέ και ελπίζω και αυτέ να κάνουν το ίδιο, να συμπεριλάβουν εμά δηλαδή αν ασχοληθούν δεν ξέρω, με την ασφάλεια ας πούμε των εξεδρών. Να δώσω ένα παράδειγμα. Και βεβαίως σωστό είναι να επισημαίνουμε την περιβαλλοντική πτυχή, την αηφορία και την αποτελεσματικότητα του κλάδου και οι προδιαγραφές ασφαλείας και η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, γιατί δεν είμαι πεπισμένος συνάδελφοι πως η συνεργασία στην θαλάσσια πολιτική μεταξύ κρατών μελών είναι τόσο καλή όσο θα μπορούσε να είναι. Υπάρχει αυτή η σκέψη του στυλ αυτά είναι τα δικά μας ύδατα, αυτή είναι η δική μας επικράτεια και ε, σε αυτό θα επιμείνουμε. Οπότε πρέπει εδώ η Επιτροπή και η Κομισιόν να προσπαθήσουν να σπάσουν αυτά τα εθνικά αν θέλετε τείχη που υπάρχουν όταν μιλάμε για τις θαλάσσιες μεταφορές. Ανέφερα την πετρελαιοκυλίδα που είναι το ζήτημα της ημέρας. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την θαλάσσια πολιτική που δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε. Υπάρχει ε, περιβαλλοντικός αντίκτυπος και για να πούμε και τα της ΕΜΣΑ η ΕΜΣΑ πράγματι παρακολουθεί τα πλοία εκείνα τα οποία καθαρίζουν ε, τις δεξαμενές τους στην θάλασσα. Χρειαζόμαστε επιτήρηση εκεί. Υπάρχει το ζήτημα της πειρατείας. Πριν από έξι μήνες, συνάδελφοι, το ζήτημα ήταν η πειρατεία. Το κοινοβούλιο απαιτούσε δράση για την πειρατεία. Τώρα απαιτούμε δράση για τις εξέδρες πετρελαίου. Ε, πρέπει να είμαστε συνεπείς και να θυμόμαστε το τι ζητήσαμε και σε προηγούμενες ε, συζητήσεις και να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση σε οποιαδήποτε ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Θυμάστε την έκθεση του Ρόμπερτ Evans για την διάλυση των πλοίων και τις ε, συνθήκες που επικρατούν στο Μπαγκλαντές. Οπότε όταν μιλάμε για ολοκληρωμένη ε, θαλάσσια πολιτική και εγώ Πιστέψτε με. Είναι τεράστιο θέμα και ένα τεράστιο κουτί αυτό το οποίο ανοίγουμε. αλλά νομίζω πως ε, εδώ πέρα υπάρχει δυνατότητα όχι μόνο στον τομέα της ε, ναυπήγησης και της διάλυσης των πλοίων. Θέλω να το δει αυτό και η κυρία Μάισνερ μπορούμε να διαλύζουμε τα πλοία με σωστό τρόπο, περιβαλλοντικά σωστό και ασφαλή, σε αντίθεση με κάποιους ε, πλειοκτήτες που τα πετάνε, προσαράζουν στις ακτές του Μπαγκλαντές και τα διαλύουν, πλοία, ε, τα διαλύουν παιδιά μετά. Η κυρία Γιάλα Σέντερ ανέφερε το ζήτημα των ε, ναυτικών και την δυσκολία του να βρούμε Ευρωπαίους ναυτικούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι θεμητό ε, ζήτημα, πράγματι. Γνωρίζω πως η Επιτροπή Απασχόλησης εξετάζει το ζήτημα των μη Ευρωπαίων ναυτικών που απασχολούνται σε ευρωπαϊκά πλοία, ειδικά τα ferry που ε, ε, δεν φεύγουν από το πλοίο επί μήνες. Πρέπει λοιπόν να δούμε πιο σοβαρά την δομή της απασχόλησης στον θαλάσσιο τομέα. Γιατί όπως είπε η κυρία Γιάλα, οι καπετάνιοι δεν είναι το πρόβλημα ε, και οι ε, Ευρωπαίοι πολίτες. Θα συμπεριλάβω εδώ πέρα και την Κροατία γιατί φαίνεται πως όλοι οι καπετάνιοι είναι Κροάτες τελευταία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στην Ευρώπη υπάρχουν καλά εκπαιδευμένοι άνθρωποι. Δεν το αμφισβητώ αυτό. Το πρόβλημα είναι το κατώτερο πλήρωμα. Και πώς θα γίνει η ναυτιλία πιο ελκυστική για τους Ευρωπαίους πολίτες και πώς θα απασχοληθούν στον ε, τομέα αυτόν. Ο κύριος Τέιλορ ανέφερε προς, ε, προέρχεται από την νότια ακτή. Εγώ Είμαι, κατάγομαι από το, μια περιοχή κοντά στο λιμάνι του Λίβερπουλ. Με μεγάλη ναυτική παράδοση. Τα παιδιά τελείωναν το σχολείο και πήγαιναν στο εμπορικό ναυτικό. Δεν γίνεται πια αυτό το πράγμα. Είναι θλιβερό. Ο κύριος Κουμουτσάκος μου άρεσε η τελευταία του παρέμβαση. Ε, δεν είμαι τόσο σίγουρος για την πρώτη. Γιατί δεν είμαι τόσο σίγουρος για την ανάπτυξη του παράκτιου τουρισμού. Ε, Βεβαίω ενδιαφέρον είναι πω προέρχεται από την Κρήτη η κυρία Επίτροπο, ένα από τα αγαπημένα μου νησιά που έχει και το καλύτερο ελαιόλαδο στον κόσμο και δεν είμαι σίγουρο εάν θα έπρεπε να προσπαθούμε να αναπτύξουμε τον παράκτιο τουρισμό. Θυμάμαι όταν ήταν και ο κύριο Σταγιάν εδώ πέρα, του είπαμε πω πρέπει να αναπτύξουμε εναλλακτικό σχέδιο τουρισμού, το οποίο θα είναι πιο αηφόρο και οικονομικά και περιβαλλοντικά. Και αυτό σημαίνει να αναπτύξουμε τον τουρισμό σε άλλες περιοχές. Ε, εκτός, να πάνε και αλλού, εκτός από τις παραλίες. Γιατί η τουριστική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπαγορεύεται από τις παραλίες και τα βουνά. Και υπάρχει και αυτή η υπερβολική ανάπτυξη που ανέφεραν οι πράσινοι, επειδή ακριβώς όλοι πηγαίνουν σε αυτόν τον τουρισμό. Εγώ δεν λέω να τα αγνοήσουμε. Αυτό το οποίο είπαμε στον κύριο Ταγιάννη είναι πως πρέπει να δούμε πιο αηφόρες μορφές τουρισμού. Και χρησιμοποίησαμε το παράδειγμα της βιομηχανικής κληρονομιάς, τουρισμό ηλικιωμένων κτλ. κτλ. το, το ειδικό καθεστώ τη Μεσογείου. Εγώ θα ήθελα να δω ειδικό καθεστώ για όλα τα ύδατα τη Ένωση. Βεβαίω οι συνάδελφοι από τη Μεσόγειο μπορούν να πούν ε, για τη Μεσόγειο, αλλά και η κυρία Τικάου μπορεί να μα πει βεβαίω πω η Μαύρη Θάλασσα θα πρέπει να ε, είναι εκεί που πρέπει να δώσουμε βάρος, όπως και εγώ μπορώ να σας πω πως η θάλασσα της Ιρλανδίας ε, πρέπει να αποτελέσει το βάρος τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό δεν μα οδηγεί πουθενά. Πρέπει να δούμε τη θαλάσσια πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και νομίζω πω η κυρία Μάισνερ πραγματικά συνεχίζει ε, τη δουλειά του Βίλι Πίτσικ και έχουμε προχωρήσει τώρα στο να δούμε τα πράγματα ευρύτερα. Και νομίζω πως ε, έτσι πρέπει να κινηθούμε. Με συγχωρείτε αν κάνω κήρυγμα, μια ερώτηση για την κυρία Επίτροπο και δεν ξέρω, κυρία Μάισνερ, να το αναφέρετε στην έκθεσή σας. Δεν ξέρω ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας. Δεν ξέρω πού βρισκόμαστε με το καθεστώς της Ένωσης στον οργανισμό. Γιατί σαφώς βεβαίως θα παλέψουν με νύχια και με δόντια τα κράτη-μέλη να κρατήσουν τη θέση τους. Αλλά εάν είναι να είμαστε επιτυχοί σε μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική μεταφορών για την Ένωση, πρέπει να ορίσουμε ποιος είναι ο ρόλος της Ένωσης στον διεθνή φορέα που εφαρμόζει αυτά τα πράγματα. Έστω και κάπως αργά βεβαίως όπως κινείται ο Διεθνής Οργανισμός Δαυτιλίας. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν την άποψη. Σκοπεύω να ακούσουμε την κυρία Επίτροπο να απαντήσει και τις 45 εκατομμύρια ερωτήσεις και μετά θα συνοψίσει η συγκεκριά, αν συμφωνείτε. Κύριε Επιτροπέ, έχει τον λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Φυσικά δεν είμαι τόσο φιλάδοξη ώστε να απαντήσω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ. Λίγο ελληνικά, λίγο. Θα ήθελα πρώτα να σας ευχαριστήσω όλους για την ε, πολύ καλή παραγωγική και δημιουργική συζήτηση. Ε, πραγματικά η πολιτική μας για τη θάλασσα είναι, η ολοκληρωμένη μας πολιτική για τη θάλασσα είναι μια νέα πολιτική. Αλλά όπως και εσείς ε, κύριε Πρόεδρε πολύ σωστά είπατε στην παρέμβασή σας και όπως και ο κύριος Κουμουτσάκος είχε την καλοσύνη να θυμίσει, δεν αποφασίζουμε τώρα για το αν χρειαζόμαστε αυτή την πολιτική. Το έχουμε ήδη αποφασίσει. Και αναφέρομαι σε αποφάσεις και της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπου με σαφήνεια διατυπώνεται η ανάγκη να προχωρήσουμε σε μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και να αξιοποιήσουμε τα ωφέλη που θα προκύψουν από τη συνεργασία όλων μας. Ε, το λέω αυτό, το διευκρινίζω απέναντι και στον κύριο στα όσα επισήμανε ο κύριος Πασκουάλ. Είχαμε συζητήσει παρόμοια ζητήματα όταν πράγματι στην ακρόασή μου και είχα παρακολουθήσει τις ανησυχίες του Θέλω όμως να του θυμίσω ότι είμαι επίτροπος, όχι όπως είπε Commissioner for Fisheries and Some Other Affairs. Ε, ε, I would like to remind to him... Θα ήθελα να του θυμίσω ότι είμαι επίτροπος για τα θαλάσσια θέματα και την αλληλεία, αυτό είναι το, αυτή είναι η θέση μου, είναι, γι' αυτό το πράγμα έδωσα όρκο και σκοπεύω να ασκήσω τις ε, δραστηριότητές μου και τις αρμοδιότητές μου και είμαι έτοιμη να δεχτώ και κριτική και από εσά ακόμη. Έχω δεχθεί εξάλλου κριτικές κατά το τελευταίο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων για την απόφαση προώθησης των θαλάσσιων υποθέσεων. Πρέπει λοιπόν να να καταβάλω ακόμα πιο σκληρές προσπάθειες. Το λέω αυτό για να διαλύσω την όποια σύγχυση, όπως είπατε. Εδώ δεν μιλούμε για σύγχυση, μιλούμε για συντονισμό. Και θα ήθελα να τονίσω και να πω ότι η έκθεση της κυρίας Μάισνερ είναι ένα εξαίρετο παράδειγμα για το τι μπορεί να επιτύχει ο συντονισμός. Να τονίσω επίσης ότι αυτό είναι ένα βήμα παραπέρα και περί αυτού πρόκειται η ενοποιημένη, η ολοκληρωμένη προσέγγιση προσπαθεί να καλύψει ακριβώς όλα τα θέματα. Αντί λοιπόν να προσπαθούμε ποιος είναι αρμόδιος γιατί, ε, ε, προσπαθούμε να συνεργαστούμε και να αποδώσουμε. Αυτή είναι η πρόθεσή μου. Ήθελα να σας πω ότι αυτό που, αυτό που είπα και στην ε, πρώτη παρέμβασή μου, να μιλήσω δηλαδή για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ήδη στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Έχουμε ήδη συζητήσει εκτεταμένα και συμφωνήσει με τους άλλους επιτρόπους και με, τα, με τους Τατζάνι, Ποτότσνικ, Κάλλας, με όλους έχουμε συζητήσει εκτενώς και συμφωνήσει και όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ελπίζω λοιπόν ότι και η δική σας επιτροπή θα προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση και ομολογώ ότι ο πρόεδρος εδώ διευκόλυνε και την δική μου ζωή με αυτά που είπε. Επί της ουσίας, για το θέμα της διακυβέρνησης, χαίρομαι πάρα πολύ που όλοι ασχολούνται με το πρόβλημα αυτό και συμφωνώ με τις ανησυχίες σας ο κύριος Κουμουτσάκος, αναφέρθηκε ο κύριος Δανέλης, οι εκπρόσωποι των, του, εκπρόσωπος των Σοσιαλιστικού Κόμματος, μετά την τελευταία απόφαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων κάποια πρόοδο σημειώθηκε. Για να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας, πιστεύω ότι ο λόγος που δεν είχε επιτευχθεί μέχρι στιγμή, καθόλου πρόοδο, είναι ο ίδιος λόγος τον οποίο συζητούμε και εμείς τώρα εδώ. Είναι όλα αυτά τα θέματα για τη σύγχυση αρμοδιοτήτων, ποιος είναι υπεύθυνο για τα θαλάσσια πράγματα, ποιος είναι ο αρμόδιος υπουργός, στον οποίο πρέπει να απευθυνθούμε κτλ. κτλ. Τώρα όμως νομίζω ότι έχουμε λάβει πια την πολιτική απόφαση. Ήδη το έχω κουβεντιάσει με πολλά κράτη-μέλη και ελπίζω ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε ένα δίκτυο σε υπουργικό επίπεδο ένα καλό δίκτυο για να εφαρμόσουμε τις πολιτικές μας αλλά είμαι πολύ ευτυχής που άκουσα τις ανησυχίες σας και με χαρά μου θα τις ε, μεταβιβάσω, θα τις διαβιβάσω στο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αφήσουμε πια τα λόγια και να προχωρήσουμε σε αποτελέσματα. Τώρα, για τη γαλάζια ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης. Ε, ναι, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε καινοτομία στις πολιτικές μας, το είπε η κυρία Μάισνερ. αυτό με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε είναι τι πρέπει να κάνουμε για να προσελκύσουμε νέα άτομα σε αυτές τις δουλειές, σε αυτά τα επαγγέλματα. Έχω συζητήσει το ζήτημα με τον Επιτροπό Άντορ που είναι υπεύθυνο για την απασχόληση και αυτό που σκοπεύουμε να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε τις συνθήκες, τις συνθήκες ασφάλειας, τις, ε, τις αμοιβέ των ναυτικών, και, στην αυτιλία και στι θαλάσσιε μεταφορές και στην αλληλεία. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Και το λέω γιατί δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά ίσως πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι πολλά κράτη-μέλη, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα κράτη-μέλη δεν έχουν επικυρώσει ακόμα, δεν έχουν επικυρώσει ακόμα τις συμβάσεις του Διεθνού Οργανισμού Απασχόλησης για τους μισθούς, για τις αμοιβέ, για τις συνθήκες εργασίας των ναυτικών και γενικά των εργαζόμενων στη θάλασσα, για την ασφάλεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά πάνω σε αυτό. Ε, γιατί ακριβώς... Επίσης και για το Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας πολλές από τις συνθήκες και τις συμβάσεις του δεν έχουν επικυρωθεί από κράτη-μέλη. Πρέπει να πω ότι εργαζόμαστε πάνω σε αυτό Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας και τον ε, πρόεδρο του οργανισμού, ίσως και να έρθει σύντομα στις Βρυξέλλες, αλλά αυτό που μπορώ να πω προς το παρόν είναι ότι προσπαθούμε να έχουμε καθιστός παρατηρητή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Καλό είναι όλα τα κράτη-μέλη να έχουν κοινή θέση πάνω σε αυτό. Τι θα κάνουμε για την πλέον ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Ε, να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, αυτό θα κάνουμε και γι' αυτό αναφέρθηκα και σε μια μελέτη που έχουμε αναθέσει για όλα τα σενάρια, τα πιθανά σενάρια και τις δυνατότητες βελτίωσης των συνθήκων απασχόλησης στον τομέα αυτό. Τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης αυτής είναι πολύ ενθαρρυντικά, γιατί μας δείχνουν ότι στον τομέα αυτό και ενώ στον τομέα της θάλασσας γενικά, στο θαλάσσιο τομέα γενικά, έχουμε πολύ περισσότερες δυνατότητες από τις δυνατότητες που έχουμε γενικά στον εργασιακό τομέα. Πρέπει λοιπόν να υποφεληθούμε αυτής της κατάστασης. Αναφερόντας τον κύριο Κάντσιαν που, ήταν πολύ απασχολημέ... που τον ανησυχούν πολύ τα αποτελέσματα, μπορώ να του πω ότι έχουμε αποτελέσματα, μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Φυσικά δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε όλες τις επενδύσεις και όλες τις πρωτοβουλίες με τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας, γιατί δεν είναι και τόσα πολλά. Αλλά 50 εκατομμύρια είναι απλώς η αρχή. Και εγώ αναμένω πραγματικά τη συνεργασία σας για να επιτύχουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών προοπτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ένωσης γενικότερα. Και αυτό με φέρνει στο τελευταία μου παρατήρηση. Πολλοί από εσά αναφέρατε την καταστροφή στον κόλπο του Μεξικού. Πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό και το κύριο θέμα που εγείρει αυτή η καταστροφή, δύο θέματα είναι. Ένα είναι ο εθισμός, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πετρέλαιο. Έχουμε εδώ ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η εξάρτησή μας από το πετρέλαιο. Πρέπει να αναπτύξουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε ήδη μερικά πολύ καλά αποτελέσματα σε μελέτες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, που προέρχονται από τη θάλασσα. Ε, συνεργαζόμαστε με τον κύριο Έρντιγκερ πάνω σε αυτό. Δεν είναι πολύ γνωστές οι πηγές ενέργειας. Αναφέρω το αιωλικό πρόγραμμα, το οποίο φυσικά το ξέρουν όλοι. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχει το θέμα της ε, παλυριακής ενέργειας, της ενέργειας από την ε, παλύρια από τον ε, κυματισμό, από, από, το θερμικό δυναμικό της θάλασσας. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές πρόπτικες. Πρέπει να επενδύσουμε στην τεχνολογία και να την εκμεταλλευτούμε. Η πρώτη λοιπόν πρόκληση που εγείρει η καταστροφή στο Μεξικό είναι αυτή η εξάρτησή μας από το πετρέλαιο. Η δεύτερη πρόκληση είναι η προστασία του περιβάλλοντος σε περιπτώσεις τέτοιων ατυχημάτων. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ασχολείται με το θέμα και σύντομα θα έχουμε μια πρωτοβουλία. Με όλους τους επιτρόπους, την κυρία Ρέντιγκερ, ε, τον κύριο Ποτότσνικ, όλοι, όλοι οι επίτροποι θα συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Πιστεύω ότι ακόμα και ο πρόεδρος Μπαρόσο θα συντηρήξει αυτή την πρωτοβουλία, θα συμμετέχει με τα χαρά μου θα μεταφέρω το μήνυμά σα προς την Επιτροπή ότι πρέπει να δράσουμε, ότι πρέπει να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένε Πολιτείε, όπως ανέφερε και κάποιος Ευρωβουλευτής. Πράγματι πρέπει να συνεργαστούμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε και να μάθουμε τα μαθήματά μας από αυτήν την καταστροφή γιατί ήδη μα έχει διδάξει πολλά πράγματα. Εν κατακλείδη θα ήθελα να, ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω όλους για τις παρεμβάσεις σας. προσπαθώ να καταγράψω όλες τις προτάσεις σας και θα ήθελα να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι Καθόλου δεν προσπαθώ να υφαρπάξω τις αρμοδιότητες άλλων επιτρόπων. Εγώ θέλω και επιζητώ μόνο τη συνεργασία γιατί πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να εκπληρώσω ορθά τα καθήκοντά μου με αυτόν τον τρόπο. Και ελπίζω πραγματικά ότι θα βρω συμμάχους ε, σε αυτή μου την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Κύριε Μάισνερ επιθυμείτε να πάρετε το λόγο, να απαντήσετε σύντομα. Θα είμαι σύντομη κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω και για τα πολλά σχόλια τα οποία ακούστηκαν. Τα περισσότερα έδειξαν σαφώς πως υποστηρίζετε την κατεύθυνση την οποία ακολούθησα, αλλά να αναφερθώ σε αυτά τα οποία είπε ο κ. Ντεγκράντες Πασκουάλ, αλλά δεν είναι όλα αυτά αρμοδιότητά μου και πίστευστε με πως ε, Ξεκίνησα με το άρθρο 50 με μια ειδική περίπτωση και εγώ είμαι μια πολιτικός που ασχολείται με τις μεταφορές και λέω τώρα τι πρέπει να κάνω εδώ πέρα παρά το ότι βεβαίως είχαμε και την έκθεση Φαντάλην όπου επαναλαμβάνονται κάποια πράγματα και έλεγα να τα επαναλάβω αυτά ή να μιλήσω για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και είπα να ακολουθήσουν ολοκληρωμένη προσέγγιση και για το δίκτυο αυτό των θαλασσίων πόλων, δηλαδή, όπου συναντιόνται άνθρωποι και από τα ναυπηγεία και ε, από τον εφοπλισμό και από τον τουρισμό. Οπότε πρέπει να έχουμε πράγματι αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Και πράγματι αναρωτιέται κανείς πρέπει να μιλήσω για την έρευνα, για την προστασία του κλίματος, για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά υπάρχουν εδώ πέρα και επιτροπή ε, περιβάλλοντος η οποία όμως δεν εμπλέκεται σε αυτή την ε, έκθεση. Πού θα συζητηθεί λοιπόν αυτό το θέμα, από το σκέφτηκα πάρα πολύ και επέλεξα την προσέγγιση που θα συζητηθει λοιπον αυτο το θεμα που το σκεφτηκα Νομίζω πως ε, είναι και στο πνεύμα του Βίλι Πίτσεκ αυτό το που έχει κάνει στο παρελθόν με μια διαφορετική έτσι, κατανομή. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας λοιπόν και αναμένω να ακούσω αυτά τα οποία θα μου πείτε και σας ευχαριστώ κυρία Επιτροπέ για την παρουσία σας και για την συνεισφορά σας και για τις απαντήσεις σας. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Μάισνερ. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που προβλέπετε για την έκθεση αυτή, η προθεσμία για καταβολή τροπολογιών 9 Ιουλίου. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας το Σεπτέμβριο, θα είστε όλοι φρέσκοι από τις διακοπές σας. Να έρθετε στην Κρήτη, κύριε Πρόεδρε, λέει η Επίτροπος. Ναι, προφανώς. Και θα ψηφίσουμε στην ε, Ολομέλεια του Οκτωβρίου 2010. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την έκθεση αυτή. Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που αφιερώσετε σε εμά και για την εξαιρετική αυτή ζήτηση που είχαμε. Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους που συνέβαλαν πάρα πολύ στη συζήτηση αυτή. Και ελπίζουμε να συνεργαστούμε πολύ κοντά μαζί σας και στο εγγύς μέλλον. Και προφανώς Ελπίζουμε κάποια μέρα να πάμε στο ιστορικό πανέμορφο νησί της Κρήτης και ποιος ξέρει, ίσως να καταφέρουμε να πάρουμε και λίγο ελαιόλαδο μαζί μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Κρήτη και μ' αρέσει πάρα πολύ και το κρητικό ελαιόλαδο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας αφιερώσατε και προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστούμε. Okay, colleagues. Λοιπόν, συνάδελφοι. Νομινίκ. Πρέπει, πρέπει να συνεχίσουμε. Ε. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ΣΤΟΑ. Θα θυμάστε πως η κυρία Τικάου και ο κύριος Κόκα μας εκπροσωπούν στην δική Διοικούσα Επιτροπή. Η κυρία Τικάου λοιπόν θα αναπληρώσει τον συνάδελφο. Σίλβια λοιπόν. Έχεις τον λόγο. Α, ο κύριος Τέιλορ έφυγε. Σίλβια έχεις τον λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα σας παρουσιάσω σύντομα τις δραστηριότητες της ΣΤΟΑ που δημιουργήθηκε με απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 22 Φεβρουαρίου του 1992, απόφαση που τροποποιήθηκε με άλλες αποφάσεις στη συνέχεια. Η ΣΤΟΑ είναι η Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης των Τεχνολογικών Εναλλακτικών λύσεων που μπορούμε να έχουμε για διάφορα ζητήματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει ως ε, ρόλο να βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην υιοθέτηση συγκεκριμένων αποφάσεων που έχουν να κάνουν με επιλογή κάποιων ε, τεχνολογικών λύσεων. Η ε, λοιπόν συμβάλλει στι εργασίε των κοινοβουλευτικών επιτροπών, καθώ επίση και σε άλλου φορεί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μελέτε, ανεξάρτητε αξιολογήσει αντικτύπου και επίση διοργανώνει φόρα και συζητήσει κατά τη διάρκεια των οποίων οι πολιτικά υπεύθυνοι αλλά και οι ε, εκπρόσωποι επιστημονικών οργανώσεων αλλά και εκπρόσωποι τη κοινωνία γενικότερα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν και να συγκρίνουν τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για την κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να σας πω ότι οι δραστηριότητες της ΣΤΟΑ έχουν ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και διαφέρουν κατά αυτόν τον τρόπο από τις ερευνητικές δραστηριότητες της γραμματείας. που πολλές φορές επικεντρώνονται σε πολύ συγκεκριμένους τομείς και έχουν ένα χρονοδιάγραμμα πιο βραχυπρόθεσμο. Η ΣΤΟΑ λοιπόν δεν κάνει συγκεκριμένες μελέτες για μια συγκεκριμένη κοινοβουλευτική επιτροπή, αλλά κάνει μελέτες οι οποίες έχουν ως στόχο να καλύψουν κατά οριζόντιο τρόπο πολλές κοινοβουλευτικές επιτροπές στι ερευνητικέ ανάγκε που έχουν σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο αλλά και μακροπρόθεσμο επίπεδο. Οι μελέτες αυτές παίρνουν τη μορφή επιστημονικών αναλύσεων που γίνονται με τρόπο απόλυτα ανοιχτό χωρίς να υπάρχει καμία εμπλοκή των ενδιαφερομένων εκείνων μερών που θα μπορούσαν να περιορίσουν το πεδίο της έρευνας στα συμφέροντά τους. Επίσης, ε, τα απορίσματα της ΣΤΟΑ είναι απολύτως αντικειμενικά, δεν εκπροσωπούν απαραίτητα την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα πορίσματα αυτά έχουν την υποστήριξη ανεξάρτητων οργανισμών στον τομέα της ε, έρευνας. Οι δραστηριότητες αυτές της ΣΤΟΑ χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προπολογισμό και υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση εσωτερική Πολιτικής σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της ΣΤΟΑ. Η Επιτροπή λοιπόν ε, ΣΤΟΑ έχει 15 μέλη έναν αντιπρόεδρο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ασχολείται με τις ε, δραστηριότητες της ΣΤΟΑ, τέσσερα μέλη από την Επιτροπή Έρευνας, δύο μέλη από την Επιτροπή Απασχόλησης, δύο επίσης μέλη από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, δύο μέλη από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς, δύο μέλη από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, Συμμετέχω λοιπόν εγώ και ο Αντιπρόεδρος Κόχα και δύο μέλη από την Επιτροπή Γεωργίας. Τα μέλη της ε, ΣΤΟΑ έχουν θητεία 2,5 ετών και η θητεία τους αυτή μπορεί να ανανεωθεί. Η Επιτροπή ΣΤΟΑ συνεδριάζει στο Στρασβούργο την 5η πρωί συνήθως κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας Δυστυχώς το πρόγραμμα των συνεδριάσεών μας συμπίπτει με συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών Πολλές φορές επιμέρους ομάδες, π.χ. η ομάδα μεταφορών των σοσιαλιστών συνεδριάζει την ίδια στιγμή. Προσπαθούμε λοιπόν κάθε φορά να βρίσκουμε τους τρόπους εκείνους που επιτρέπουν σε όσο δυνατόν περισσότερα μέλη της ΣΤΟΑ να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της ΣΤΟΑ και προσπαθούμε να αποφύγουμε να συμπίπτουν λοιπόν οι συνεδριάσεις μας με συνεδριάσεις άλλων επιτροπών ή πολιτικών ομάδων. Υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια της ΣΤΟΑ που έχουν να κάνουν με τις μεταφορές η Αντιπρόεδρος Κόχο και άλλοι συνάδελφοι ασχολούνται με τα σχέδια αυτά. Στις αρχές ε, του έτους έγινε μία πρώτη συζήτηση για κάποια πιθανά σχέδια στον τομέα των μεταφορών και ε, υποβλήθηκαν ε, τρία σχέδια μελέτης και δύο επίσης σχέδια υποβλήθηκαν από μένα και από τον κύριο Ταταρέλα. Οι προτάσεις λοιπόν της Επιτροπής Μεταφορών είναι οι ακόλουθες. ηλεκτρικά συστήματα για τον τομέα των μεταφορών και της κινητικότητας της πόλης, ποιες είναι οι δυνατότητες που προβλέπονται, που μπορούν να μας δώσουν τα ηλεκτρικά ποδήλατα, τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα, η σιδηρόδρομη νέας γενιάς. Το σχέδιο αυτό λοιπόν επελέγει για να χρηματοδοτηθεί μαζί με το σχέδιο για τις οικολογικές μεταφορές και μαζί με τα σχέδια τα οποία έχουν ως στόχο να μειωθούν, να μειωθεί η χρησιμοποίηση των καυσίμων στις θαλάσσιες μεταφορές. Τα σχέδια λοιπόν αυτά τα οποία ανέφερα θα χρηματοδοτηθούν από κοινού στα πλαίσια των των περιβαλλοντικά αποτελεσματικών μεταφορών και επίσης προτείναμε μια καλύτερη αύξηση των μέτρων ασφαλείας στα αεροδρόμια. Το σχέδιο αυτό πήρε λιγότερους πόντους κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Ωστόσο, θα ενσωματωθεί στις εργασίες μας, αλλά σε μικρότερη κλίμακα. Ο κύριος Τατερέλα έκανε μία σχετική πρόταση με τίτλο «Μία νέα εποχή» όσον αφορά τις μηχανές τύπου σκάνερ, όσον αφορά δηλαδή τους αρωτές. Προβλέπεται λοιπόν να γίνει και εδώ πέρα μια έρευνα, ένα σχέδιο μικρότερης κλίμακας όμως από αυτή που αρχικά προβλεπόταν στην πρόταση. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι ε, σύντομα Οι ενδιαφερόμενοι ακόμα και αύριο το πρωί από τις 9.30 μέχρι τις 11.30 θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο που οργανώνει η ΣΤΟΑ με τον ακόλουθο τίτλο πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την, τα προβλήματα της ενέργειας κυκλοφορίας μετά την έκρηξη του ηφαιστείου. Θα υπάρχουν διάφοροι εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα μας δώσουν τη δικιά τους άποψη για το πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με την κρίση στο μέλλον κρίση δηλαδή όσον αφορά την ευαισθητική τέφρα. Επίσης, να σας πω ότι ε, στην αρχή της εντολής της ΣΤΟΑ υποβλήθηκαν 23 σχέδια προς εξέταση, προκειμένου δηλαδή να γίνουν ερευνητικά προγράμματα τρία υποστηρίχθηκαν από τους συντονιστές της Επιτροπής μας, δύο ακόμα σχέδια υπέβαλα εγώ και ο κύριος Ταταρέλα και το πρώτο σχέδιο το οποίο θα προωθηθεί από τη ΣΤΟΑ είναι το σχέδιο εκείνο που έχει να κάνει με την οικολογική αποτελεσματικότητα, όπου θα ασχοληθούμε πιο συγκεκριμένα με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά ποδήλατα και με τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μπορούμε να τροφοδοτούμε με ηλεκτρισμό τα νέα αυτά οχήματα. Θα ήθελα να ολοκληρώσω το σημείο αυτό λέγοντάς σας ότι στην είσοδο της αίθουσας μπορείτε να δείτε κάποιες δημοσιεύσεις της ΣΤΟΑ, μία περιγραφή της Επιτροπής ΣΤΟΑ, καθώς επίσης και το ενημερωτικό μας φυλάδιο, το newsletter, που θα μπορέσει να ενημερώσει τις τελειοτητές μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη σας για τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τίκαου. Ερωτήσεις, σχόλια. Ναι, ευχαριστώ. Κύριος Γκρός. Ε, ο συνάδελφος ε, Κνόχ δεν έχει φτάσει ακόμη, αλλά εν πάση περιπτώσει σας ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση και έχω δύο-τρεις πρακτικές ερωτήσεις να σας υποβάλω. Στο έγγραφο γίνεται λόγος για το μέλλον των ευρωπαϊκών μεταφορών και θα έλεγα πως προκύπτουν κάποια γενικά ερωτήματα εδώ πέρα για εμάς και τους συναδέλφους. Ποιος συντονίζει, ε, υποθέτω ότι έτσι πρέπει να γίνεται, τις διαφορετικές αυτές μελέτες που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο Κοινοβούλιο Εξονόματος ή κατ' ε, του Κοινοβουλίου είναι νομίζω σημαντικό αυτές οι πρωτοβουλίες να μην γίνονται έτσι παράλληλα γιατί βεβαίως ε, είναι και το ζήτημα το χρηματικό και όλοι ανησυχούν ε, για το ότι πρέπει να αξίζει κάτι παραπάνω από το χαρτί στο οποίο τυπώνεται η μελέτη. Να μην γίνονται δηλαδή παράλληλα μελέτες. Εσείς είπατε πως δεν γίνονται οι κατεντολήν μίας επιτροπής και κάθε ε, επιτροπή μπορεί βεβαίως να αναθέσει κάποιες μελέτες ε, μέσω της αλλά θα ήθελα να γνωρίζω γίνεται συντονισμός ή όχι. Δεύτερον, οι διαγωνισμοί πώς γίνονται, ποιος κάνει τις μελέτες, είναι πάντα προκαθορισμένα γραφεία που το κάνουν αυτό ή υπάρχει μια ειδική διαδικασία. Και τρίτον, εάν δούμε τώρα το συγκεκριμένο παράδειγμα εδώ πέρα, εντάξει, η ιδέα είναι πολύ καλή και έχει πολλές πληροφορίες, αλλά βλέπω παραδείγματο χάρη πως περιορίζεται αυτή η μελέτη στην Ουγγαρία, την Ελλάδα και τη Δανία. Οπότε το ερώτημα είναι εάν μιλάτε για τις μεταφορές, εάν εγώ ήθελα να ερευνήσω τις ε, μεταφορές μεγάλων αποστάσεων στην Ευρώπη, ποιος ορίζει ότι αυτό αφορά μόνο αυτές τις τρεις ε, χώρες. Ε? Θα ήθελα λοιπόν να απαντήσετε αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σελχαντραουή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να δώσω μέρος της απάντησης, ίσως γιατί Εγώ ήμουν μέλος του πάνελ της ε, ΣΤΟΑ, ήμουν ε, συντονιστής ε, για την έρευνα ακριβώς αυτήν πριν από πολλά χρόνια για τις μεταφορές μεγάλες αποστάσεων και να σας πω λίγο κάποια πράγματα για τους περιορισμούς της ΣΤΟΑ για το πώς ε, λαμβάνει ένα ερευνητικό Ινστιτούτο το έργο και ανεξαρτήτως από αυτό αυτό γίνεται, η επιλογή των κρατών μελών που φοράει η έρευνα γίνεται από αυτόν ο οποίος αναλαμβάνει την, ε, την ε, μελέτη. Οπότε δεν ξέρω αν γίνεται αυτό το οποίο ζητήσατε τώρα. Υπήρχε λοιπόν εδώ πέρα μία έρευνα σε τρεις φάσεις και η μελέτη για τις χώρες αποτέλεσε ένα μικρό κομμάτι στο, στο τέλος μόνο. Και εξετάσαμε μία διαφορά διαφορετικών επιλογών και το σημαντικότερο νομίζω ήταν το πρώτο κομμάτι της μελέτης όπου πανεπιστημιακοί και ερευνητικά Ινστιτούτα ε, ξεκίνησαν από κάποιες επιλογές πολιτικής ε, και μετά από αυτό βγάλαμε κάποια συμπεράσματα για τα μέτρα τα οποία έπρεπε να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τόσο αυτά μπορείτε και να διαβάσετε. Σύντομο, σύντομα τώρα, αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι πως στο Αυτό το οποίο αναμένουμε από αυτούς που είναι μέλη της ΣΤΟΑ είναι να διαλέγουν φακέλους που πρέπει να ερευνηθούν και που θα είναι σημαντικοί και θα έχουν σημασία σε δύο-τρία χρόνια γιατί μιλάμε για τέτοιες ε, προθεσμίες. Γιατί βέβαια από όταν δοθεί εντολή χρειάζεται λίγο χρόνος, πρέπει να γίνει η μελέτη και τα λοιπά. Από όταν ανατεθεί περνάνε κάτι χρόνια. Οπότε για τις αποφάσεις λαμβάνονται τώρα συμφωνώ πως ε, πραγματικά οι οικολογικές μεταφορές νομίζω μπορεί να είναι το πρώτο μεγάλο έργο, πράγματι κινητικότητα. Και έχω μια ερώτηση, μπορεί να μας απαντήσει ίσως η Σίλβια, τι ακριβώς έχετε συμφωνήσει τώρα, ποιο είναι το timing εδώ πέρα, τι μπορούμε να περιμένουμε ως αποτελέσματα, θα είναι κάποιο έγγραφο, ε, θα ακολουθήσουν και άλλες μελέτες. Και τέλος, ε, κύριε Πρόεδρε, νομίζω πως ε, όταν ε, το η ΣΤΟΑ θα αναθέσει και άλλες μελέτες του χρόνου, θα μπορούσαμε ίσως να ασχοληθούμε με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ματιέ Γκρός, δηλαδή να θέσουμε κάποιους μεσοπακροπρόθεσμους στόχους ε, το 2020, να έχουμε δηλαδή μετρήσιμους στόχους και να ερευνήσει η ΣΤΟΑ ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν σε διάφορα επίπεδα για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι αποτελεσματικά αυτή την πρόταση έχω. Τέλος, κυρία Μάισνερ, ε, σας υπενθυμίζω πως σε λίγο έχουμε και συνεδρία των συντονιστών. Ναι, κυρία Μάισνερ, δεν θα μακρηγορήσω. Κάποια πράγματα απαντήθηκαν ήδη. Εγώ θα ήθελα να γνωρίζω συγκεκριμένα πότε αναμένεται αποτελέσματα. Αυτά είναι θέματα που αφορούν και το μέλλον και παίζουν σημαντικό ρόλο στην έκθεση Γκρός και τι προγραμματίζεται. Θα ήθελα και εγώ να ξέρω το χρονοδιάγραμμα και να δούμε τι θα γίνει και στην ε, συνέχεια. Τι θα κάνουμε δηλαδή ως εφαρμογή για αυτό το πράγμα, για τις ε, μεταφορές, ε, παραδείγματος χάρη. Ευχαριστώ κυρία Σαλνόβα.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 ε, υπήρχε ένα πρόβλημα στο, στην διερμηνία. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να επαναλάβω το ερώτημα του κ. Αλχαντραουή. Πώς δοθε, δίνονται οι ε, μελέτες. Ε, είναι σκληρό να λέμε ότι μου φαίνεται ότι είναι όλο τα ίδια πανεπιστήμια. Ή ε, κατανέμονται πιο δίκαια, ας πούμε. Με κάθε σεβασμό προς την κυρία Μάισνερ, αλλά η Καλσρούη εδώ πέρα είναι συνέχεια μέσα. Οπότε πώς κατανέμονται οι μελέτες και πώς ε, τα πανεπιστήμια μας ε, μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση και να καταθέσουν μια προσφορά για την στο Σιλβία. Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλους. Καταρχήν, όσο αφορά την ερώτηση του κυρίου Γκρός, ε, δυστυχώς υπάρχει και ένα τεχνικό πρόβλημα. Ένας, ε, ένας βουλευτής μπορεί να αποστείλει σε μια επιτροπή ΣΤΟΑ αίτηση για κάποιο μελέτη, κάποιο σχέδιο. Στη διάρκεια του χρόνου ένας βουλευτής ή μια επιτροπή κοινοβουλευτική μπορεί εκ νέου να υποβάλει αίτημα για κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα. Λαμβάνουμε πολλές αιτήσει, πολλά αιτήματα. Ο προϋπολογισμός μας είναι περιορισμένος. Γίνεται ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Επιτροπής ΣΤΟΑ και... Ε, όσα ερευνητικά σχέδια συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία, χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό μας. Επίσης έχουμε και κάποιες τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ανάθεση των ε, μελετών. Για το άρθρο του κανονισμού της ΣΤΟΑ, σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό και τις εκτελεστικές πράξεις, ε, οι στρατηγικές επιλογές, τα θέματα αποφασίζονται και ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες και ανάλογα με την ψηφοφορία λοιπόν επιλέγονται τα προγράμματα και ο, συντονιστή, ο αρμόδιος συντονιστής των πιστώσεων μετά από αίτηση της Επιτροπής πρέπει να ακολουθήσει της, ε, τη διαδικασία ενός δημόσιου διαγωνισμού. Κάθε ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πολλές ερευνητικές υπηρεσίες σε πολλά κράτη-μέλη. Υπάρχει μια σειρά κριτηρίων που πρέπει να ικανοποιούνται. μεταξύ των οποίων η παρουσίαση των αποτελεσμάτων κατά τρόπο που να είναι κατανοητός από όλους υπάρχει άλλος εξωτερικός αξιολογητής, αξιολογητής που δεν, έχει, δεν βρίσκεται σε σχέση με τη ΣΤΟΑ, δεν έχει αναλάβει κανένα ερευνητικό πρόγραμμα από την ΣΤΟΑ. Συνήθως ε, οι σχετικές μελέτες διακρίνονται από υψηλή επιστημονική ποιότητα. Ελπίζω ότι απάντησα στα, στις ερωτήσεις ε, στις ερωτήσει σας. Τα ερευνητικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια που ενδιαφέρονται μπορούν να συμμετέχουν είτε για να τους προ σχέδια ε, σε αυτά ατομικά, είτε μπορούν να σχηματίσουν ε, κοινοπραξίες για να συμμετάσχουν στους δημόσιους διαγωνισμούς. Στην κυρία Μέιστνερ, υπάρχουν ευραχυπρόθεσμα σχέδια ε, τριών με εννέα μηνών και μεσοπρόθεσμα σχέδια καθώς και μακροπρόθεσμα σχέδια που μπορεί να εκτείνονται σε τρία χρόνια. Το σχέδιο για τις μεταφορές θα είναι μακροπρόθεσμο, θα ξεκινήσει πολύ σύντομα, θα είναι μακροπρόθεσμο όπως είπα και θα λαμβάνει υπόψη ε, όλα αυτά που είπε ο κύριος Καντράουι. Δηλαδή θα δούμε κατά πόσο μεταξύ των τεχνικών προδιαγραφών ποιες από τις τεχνικές προδιαγραφές ανταποκρίνονται στο πνεύμα της έκθεσης του κυρίου Γκρός και μπορεί να περιλαμβάνουν συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους, στόχους που έχουν αποφασιστεί από την Επιτροπή Μεταφορών. Πιστεύω ότι έχω απαντήσει πάνω κάτω Λοιπόν, ποιοι αναλαμβάνουν αυτές τις μελέτες, ερευνητικά ιδρύματα ή πανεπιστήμια ή κοινοπραξίες μεταξύ αυτών. Οι επιτροπές και οι βουλευτές μπορούν πάντοτε να υποβάλουν αιτήματα, αλλά όπως σας είπα, η Επιτροπή ΣΤΟΑ δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει παρά μόνο οριζόντιες μελέτες. Αν λοιπόν ζητούμε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που να εντάσσεται αυστηρά μόνο στο πλαίσιο των μεταφορών, η ΣΤΟΑ δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα τέτοιο σχέδιο. Ελπίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις σας. Αν όχι, παραμένω στην διάθεσή σας. Αν έχετε και άλλες ερωτήσεις, ευχαρίστως να τις απαντήσω. Σας προτείνω να σας ενημερώνουμε περιοδικά, είτε μεμονωμένα, είτε να ενημερώνουμε όλη την Επιτροπή, έτσι ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε τα ερευνητικά σχέδια που έχουν ενδιαφέρον για την Επιτροπή σας. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ, κυρία Τίκαου. Ευχαριστώ και τον κύριο Κοκ. Και τους δύο σας ευχαριστώ. Το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι τα διάφορα. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο θέμα. Σας υπενθυμίζω την ημερομηνία και τον τόπο της επόμενης συνεδρίασης. Βρυξέλλες, Δευτέρα, 12 Ιουλίου, στις 3 η ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσει τώρα η συνεδρίαση των συντονιστών. Οπότε λύεται η συνεδρίαση. Ευχαριστώ.